οι συναδέλφισες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι ευχάριστο που παρά το γεγονό ότι ξεκινάμε στις 2.30 έχετε έρθει αρκετοί και επειδή μα περιορίζει πάντα ο χρόνο, θα περάσουμε κατευθείαν στη μερίσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε την έγκριση τη μερίσια διάταξη. Μπορούμε να πούμε ότι συμφωνείτε όλοι. Προφανώς, οπότε στην τρέχουσα μορφή τη μερίσιας διάταξη εγκρίνεται και προχωράω στι ανακοινώσει της Προέδρου. Διερμηνία. Έχουμε τις ακόλουθες γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγαρικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα. Η συνεδρίαση αυτή είναι web streamed και θα ήθελα να σημίσω την αυτόματη διαδικασία που ισχύει και να σας παρακαλέσω και στις ομάδες σας να ε, κερδίσετε την υποστήριξη για την ε, αυτόματη ε, έγκριση των ψηφισμών που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση Θα ήταν πολύ καλό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το ψήφισμα. Θα είναι αργά να αποφασίσουμε μετά αν ήδη τα έχει αποφασίσει πρώτα το Συμβούλιο. Αυτό ε, για να βοηθείτε μπορείτε να απευθύνετε στους ε, συντονιστές με email και να επισημάνετε φυσικά τη σοβαρότητα του θέματος ε, στις πολιτικές σας ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Κλείνοντας αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας θυμίσω την ε, ε, την ε, συνεδρίαση στις 20 Νοεμβρίου. Είναι το έτος πολιτισμικής κληρονομιάς 19 και 20 Νοεμβρίου απέχουν λίγο ακόμα, αλλά θα ήθελα από σήμερα να σας ε, θυμίσω ότι είναι σημαντικές ημερομηνίε. Και αναφερθήκαμε σε αυτό και στην προηγούμενη συνεδρίαση με τους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και συμφωνήσαμε ότι πολλά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήταν ε, δεν με παρόντα επισκιάστηκαν από την απουσίαζε αντίστοιχη παρουσία από το Ευρωκοινοβούλιο. Σας παρακαλώ λοιπόν τις ημερομηνίε αυτές, 19 και 20 Νοεμβρίου, να τις σημειώσετε στο ημερολόγιο σας. Το Save the Date ε, το λάβετε ήδη πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και την οριστική πρόσκληση την έστειλα την προηγούμενη εβδομάδα στους ε, συναδέλφους. Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία και προσδοκώ μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια περνάμε στο σημείο 3 γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ESF+. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι πολύ κοντά στις 27 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα. Γνωρίζετε όμως ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί υπάρχουν διάφορες νομοδοτήσεις και διαφορετικές διάφορες επιτροπές και αυτό μας ε, θέτει υποπίεση. Παραλαμβάνω 27 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα και εφόσον είμαι εγώ η συγγήτρια θα ξεκινήσω με μια εισαγωγή. Το σχέδιο γνωμοδότησης το έστειλε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ πρέπει να υπάρχει σε όλες τις ε, γλώσσες. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας, σύμφωνα με το άρθρο 54C, ε, εμπλέκεται. Έχουμε λοιπόν μια καλή ευκαιρία η θέση μας να μπορέσει να συμπεριληφθεί στην ε, τελική έκθεση της Επιτροπής Επιτροπής. Αναμένω λοιπόν στις επόμενες εβδομάδες να συζητήσουμε αυτό το φάκελο και να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχει εδώ και 60 χρόνια και είναι το πιο σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια άμεση επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ανθρώπους και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να συνδυαστεί με ένα ανανεωμένο κοινωνικό ταμείο, το ESF+, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω. Η πρόταση κανονισμού της 23 Μαΐου για το ESF Plus ε, προτείνει κάποιες ε, νέες, κάποιες καινοτομίες. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον το ESF Plus θα είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο που θα στηρίξει τον πυλώνα της, ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, υψηλού επίπεδου απασχόληση, προστασίας, κοινωνική προστασίας, εργαζομένων με υψηλά προσόντα, ισότητα ευκαιριών, δίκαιες συνθήκες ε, εργασίας και υψηλό επίπεδο υγειονομική περίθαλψη. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, λοιπόν, όπω βλέπετε μελλοντικά. Στο πλαίσιο του ESF θα ενταχθούν ε, διάφορα προγράμματα τα οποία θα είναι πιο ευέλικτα και πιο απλουστευμένα. Αυτό που είχαμε προηγουμένως με το πρόγραμμα Erasmus Plus έχει να κάνει με το ESF, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για ε, περιθωριοποιημένα άτομα και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Τρει είναι οι στόχοι. Βελτίωση τη συνοχή και των συνεργειών μεταξύ συμπληρωματικών ευρωπαϊκών μέσων που θα υποστηρίξουν ε, τους ανθρώπους και θα βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Η περισσότερη ευελιξία και δυνατότητα για μια καλύτερη αντίδραση των ταμείων στον κύκλο των πολιτικών ε, ε, και οικονομικών αποφάσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, την απλούστευση του προγραμματισμού και της διοίκησης, ώστε το διοικητικό άχθος να μειωθεί. Μια περαιτέρω σημαντική αλλαγή είναι η σύνδεση του ESF Plus με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καθώς και με τις καταχώρες συστάσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει στο μέλλον να έχουν ε, ε, τις απαραίτητους πόρους για την ε, αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή σύμφωνα με τις καταχώρες συστάσεις. Το πώς θα εφαρμοστεί αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει ακόμα να αποσαφινιστεί Η πρόταση της Επιτροπής έχει σίγουρα τα δυνατά της σημεία, αλλά σε κάποια σημεία ε, δεν ανταποκρίνει τουλάχιστον στις δικές μου προσδοκίες. Γι' αυτό έχω προτείνει 29 τροπολογίες. Από τη δικιά μου οπτική υπονομεύει η σύνδεση του ESF Plus και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τις καταχώρες στάσεις στη φύση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και πιο συγκεκριμένα την διατήρηση τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό το λόγο έχω προτείνει κάποιε τροπολογίε σύμφωνα με τι οποίε τα κράτη-μέλη θα μπορούν εξάρτητα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τι καταχώρε συστάσει να συνεχίσουν να χρηματοδούν περιφερειακέ στρατηγικέ μέσω του ESF. Έχω και άλλες ε, προτάσει τροπολογιών για την ε, κατανομή του προπολογισμού δεν, υπάρχει, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα πρέπει να επενδύσουν τα κράτη-μέλη για την κοινωνική ε, έντοξη. Το 25% των πόρων για την ε, κοινωνική ένταξη και επιπλέον 2% για την ενίσχυση των ε, ε μειονεκτούντων ατόμων. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και προτείνω αύξηση το προπολογισμό από το 10% στο 15%. Οι χώρες που είναι ε, κάτω από το, NIT, το ποστό NIT να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα του ESF για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στις ε, περιοχές σε σχέση με αυτά που είναι πάνω από το μέσο όρο. Παράδειγμα, η Γερμανία Ε, Στο e rate είναι κάτω από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σε κάποιες περιφέρειες της Γερμανίας είναι πάνω από το μέσο όρο. Και αυτό πρέπει την Επιτροπή είναι να μην έχουν αξιώσει στα, από αυτή την περιφέρεια τη συγκεκριμένη στην Ανατολική Γερμανία για ε, τη χρηματοδότηση αυτή. Όμω πρόκειται για μια περιοχή η οποία πλήττεται από την ενεργεία των... Ε, υπάρχουν περιοχές που, έχουν πρόβλημα με την ενεργεία των νέων και γι' αυτό προτείνω και την τροπολογία. Ω ε, εισηγήτρια, ένας βασικός μου στόχος είναι να ε, εντάξει τη διάσταση της, του πολιτισμού στο τομέα της κοινωνικής ένταξης, να αυξηθεί έρθει η κινητικότητα των νέων, να αντιμετωπίσουμε την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και να αποφύγουμε και να προστέψουμε τα παιδιά από την φτώχεια. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών την έχουμε πει ήδη, αλλά θα προτείνω και άλλε στην πορεία, γιατί εξαιτία τη πίεση χρόνου ε, δεν μπόρεσα να λάβω ε, υπόψη αρκετέ πτυχέ του θέματο. Επομένω, θα προσθεθούν κάποιε ακόμα τροπολογίε που έχουν να κάνουν ε, με την εστίαση στις ε, μειονότητες, την διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ε, την εκπαίδευση στην νηπιακή και παιδική ηλικία, την καλύτερη συμπερίληψη στο πρόγραμμα Εράσμους, την απλούστευση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, δεν μα έχει εξηγήσει η Επιτροπή πώς ε, βλέπει αυτή την ε, ε διαχωρισμό μεταξύ των προγραμμάτων και επίση ο ρόλο του αθλητισμού ε, για την κοινωνική ένταξη. Όλες αυτά τα θέματα ε, μας ενδιαφέρουν πολύ και εμένα και τους συναδέλφους μα και αυτό φάνηκε στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε με την υποστήριξη της Επιτροπή Κούλ στις 4 Σεπτεμβρίου και πρέπει να, θυμηθούμε, να σας θυμίσω ότι έχουμε μία δεύτερη συνεδρίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτή την εβδομάδα. Πρόσκληση λάβατε πριν το καλοκαίρι. Θεωρούμε ότι η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ανυπομονώ να δω τη δική σας άποψη. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Επιτροπή Απασχόλησης ώστε να μπορέσουν να ε, εισρέψουν οι προτάσεις μας και στην ε, τελική, στο τελικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στους σκιώδεις ε, εισηγητές. Μόνο δύο είναι παρόντες αυτή τη στιγμή. Και θα ξεκινήσουμε την κυρία Evans. Δύο με τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Νομίζω ότι κάνατε πολύ καλές συστάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και υπάρχουν πολλά σημεία που είχα δεχτεί ιδιαίτερα τον εστιάσουμε την προσοχή μας στους νέους. Υποστηρίζω την κατανομή χρηματοδότησης, 25% κοινή χρηματοδότηση και ειδική στόχοι για, ε, για να μην υπάρχουν κοινωνικοί αποκλεισμοί. Μιλάμε για παιδιά περιθωριοποιημένους, ε, μακροχρόνια ανέργους και ούτω καθεξής. Και φυσικά και το θέμα του πολιτισμού θα πρέπει να τονιστεί. Η πρόσβαση στον πολιτισμό έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να δούμε πώς τα προγράμματα όπως το Erasmus Plus θα είναι συμπληρωματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus στην Ουαλία, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, ε, έχουμε μεγάλη χρηματοδότηση και είχαμε ιδιαίτερα επιτυχή προγράμματα. Ιδιαίτερα από μία οργάνωση γυναικών, ένα δίκτυο γυναικών για την ισότητα των δύο φύλων και βοηθήσανε χιλιάδες γυναίκες όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά να έχουν κατάρτιση, να γίνονται διευθυντικά στελέχη, να έχουν ηγετική θέση στις ομάδες και ούτω καθεξής. Επίσης, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Γι' αυτό το ESF μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό και θα ήθελα να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίλτ. Εάν επιθυμείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής με ενισχύει, διότι όπως και η πολιτική συνοχής, η πολιτική της ένταξης, ενσωμάτωσης των ε, μεταναστών περιλαμβάνεται στην κοινωνική συμπερίληψη, το κεφάλαιο τη κοινωνική συμπερίληψη, όπου υποτίθεται ότι οι χώρε μέλη θα δίνουν 25% των πόρων σε κοινή διαχείριση, πολύ περισσότερο από τα 10% που διατίθεται για την αντιμετώπιση ενεργεία των νέων. Με ενισχύει επίση διότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να κρίνει τι μεταναστευτικέ πολιτικέ των χωρών μελών και να βάζει και το χέρι τη στην τσέπη του. ήδη έχει επιπλήξει τη Γαλλία για θέματα ε, ένταξης στην αγορά εργασίας μεταναστών. Θεωρώ ότι πρόκειται για μέτρα διακριτικής θετικής μεταχείρισης. Ενώ οι στόχοι της ε, μεταναστευτικής πολιτικής πάει να τους γράψει σε πέτρα. Προσπαθεί δηλαδή να πιέσει με κάθε τρόπο η Κομισιόν χώρες όπως η Ουγγαρία, την οποία στιγματίσατε στην προηγούμενη Ολομέλεια και νομίζω ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, κοιτάζω στην αίθουσα, εάν ίσω κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ο κύριος Όφλιν. Ένα λεπτό σας παρακαλώ κύριε. Ευχαριστώ. Επισημένω στην ιδιαίτερα ε, επιδέξια διατυπωμένη εκθεσή σας κύριε Πρόεδρε βλέπω μια αδυναμία στην ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επειδή είμαι και πρώην μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Συμφωνώ με αυτό που λέτε, διότι έχω ακούσει συχνά τον κύριο Ντράγκη να μιλάει για τις αγαπημένες του διαστροτικές μεταρρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση δεν εννοούσε υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, αλλά χαμηλότερο. Δηλαδή αργότερα να παίρνει ο κόσμος σύνταξη, να μειωθούν τα διάφορα ευεργετήματα. Αυτό το σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στο κοινό νόμισμα φαίνεται να αντιβαίνει στους στόχους που έχετε καθορίσει εσείς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όχι μόνο με τις, με, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και με τις μακροοικονομικές πολιτικές τις οποίες επιβάλλει η Ένωση σε χώρες όπως η Ελλάδα και οι οποίες εγγυημένα θα αυξήσουν το επίπεδο της ανεργίας των νέων και όντως το έχουν κάνει. Δεν είναι σωστή λοιπόν η ευθυγράμμιση των πολιτικών και είναι, πρόκειται απλώς για ένα χανζαπλά στο οποίο πάμε να κολλήσουμε σε βαθιές πληγές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κώστα. Ευχαριστώ για αυτή τη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι είναι πλήρης και επίκαιρη γιατί όπως είπε και πριν αναφερόμαστε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένας βασικός πυλώνας και αυξάνεται βαθμία. Δηλαδή περνάμε στο 27% σε σχέση με το 23% που προϋπήρχε και περιλαμβάνει και τα τέσσερα άλλα βασικά ταμεία. Ελπίζουμε αυτό να μην προδικάσει την ιδιαιτερότητα αυτών των ε, ταμείων και γι' αυτό κάνω μία σύσταση για αυτή την ιδιαιτερότητα γιατί στον, στον προηγούμενο προϋπολογισμό φοβηθήκαμε ότι ο κανονισμός που ισχύει για το ΕΚΤ θα ισχύσει και για, για το Ταμείο για τους πλέον ενδεείς. Και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μεταξύ των ε, νέων κριτηρίων κατανομής εντάσσονται και αυτά τα NEET, δηλαδή που αφορούν ε, τομείς εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Ε, πρότεινες αυτή ε, η χρηματοδότηση να προβλέπει μία ποσόστοση για το ΝΙΤ και για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υψηλή χρηματοδότηση. Ε, είναι μία ε, ερώτηση και θέλω μία απάντηση. Δεν είμαστε και τόσο πολύ σήμερα. Αυτή η ποσόστοση που ισχύει για τα κράτη-μέλη που δεν ε, συμπεριλαμβάνονται, όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιφέρειες γιατί έχουν άλλο επίπεδο net, ε, θα πρέπει να έχουν αυτές τις χορηγίες εκτός των περιφερειακών που ήδη, όπου ήδη υπάρχει ειδική χρηματοδότηση. Πριν να επισέλθω στο ερώτημά σας, στρέφω τα βλέμματα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν ίσως θέλει κάποια εκπρόσωπό της να παρέμβει. Όχι. Ωραία. Να απαντήσω τότε στην ερώτησή σας. Στην πρόταση πρόκειται περί του εξής. Ορισμένα κονδύλια θα μπορούν να διατίθεται ιδίω για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μόνο όταν η ποσόστοση NEET βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ένωσης. Και NEET σημαίνει πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση ή σε απασχόληση ή σε κατάρτιση κλπ. Όμως υπάρχουν ορισμένε χώρες που είναι πάνω μεν από τον μέσον όρο, δηλαδή είναι κάτω από τον μέσον όρο σε ό,τι αφορά τα άτομα νιτ, ορισμένε περιφερειέ τη όμω είναι πάνω από τον μέσον όρο σε, αφορά, σε άτομα νιΤ. Και γι' αυτό εκεί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, μόνο και μόνο, επειδή η χώρα μέλος είναι κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή έχει λιγότερα άτομα από το μέσο όρο σε κατάσταση νιτ. οι περιφέρειες εκείνες οι οποίες ωστόσο έχουν παραπάνω από την ποσόστοση να μην λαμβάνουν κονδύλια για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων. Και έτσι, για να μπορέσει να υπάρξει μια περιφερική εξισορρόπηση και μέσα στις ίδιες τις χώρες μέλη. Και να μπορούμε να πούμε ότι οι χώρες μέλη που, ε, πλήγονται, που πλήττονται συγγνώμη, ιδιαίτερα από ανεργία των νέων να μπορούν να λαμβάνουν τέτοια μέτρα και ιδίως ξαναλέω όταν η, εθνική ποσόστοση βρίσκεται κάτω από τον μείζον όρο της Ένωσης. Νομίζω ότι κάποτε τα ε, διάφορα κοινωνικά ταμεία φτιάχτηκαν ακριβώς και για αυτό το λόγο, για να υπάρξει και να αποκατασταθεί μια ε, ισορροπία μεταξύ των περιφερειών. Χτες όμως ε, συζητήθηκε αυτό το θέμα για την κατάσταση της Ιταλίας, όπου ο Βοράς βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τον Νότο. Και πρόκειται για μία χώρα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ε, ε, θύλακες με μεγάλη ανομοιογένεια και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επικρατήσει η κοινωνική δικαιοσύνη παντού. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αναμένω με ενδιαφέρον ε, τις ε, ενδεχόμενες τροπολογίες σας και όπως είπα τούτη εδώ τη βδομάδα θα γίνει άλλη μια συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών και ίσως προκύψουν κάποιες εισρωές από κάποιες πλευρές, κάποια input δηλαδή. Υπενθυμίζω προθεσμία εκατάθεση τροπολογιών η 27η Σεπτεμβρίου ε, το απόγευμα και 8 Νοεμβρίου θα ε, γίνει η ε, ψηφοφορία εδώ σε Παριμήν και τέλη Νοεμβρίου η Επιτροπή Απασχόλησης. δηλαδή σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και Έρχομαι στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το υπαρθμόν 4, όπου προβλέπεται ψηφοφορία για γνωμοδότηση της κυρίας Μποσκόρ για ελάχιστους κανόνες υπέρ μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας και επιθυμώ να ε, ρωτήσω την κυρία Μποσκόρ αν έχει να πει κάτι ή αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Καλώς, μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία, όπως ε, μου δείχνει η κυρία Μποσκόρ. Μια στιγμή να βγάλω και εγώ την κάρτα ψηφοφορίας. Με κυρια βοσκορ μια στιγμή να την βρω στην τσάντα μου. Έχετε όλες και όλες τις κάρτες σας. Ωραία. Μπορούμε να αρχίσουμε με την, με την συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαρχούν 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές Α, νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απερίφη όμως 7 προς 9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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να επαληθεύσουμε 44 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απερίφθη 10 κατά 6 υπέρ δύσκολο να το δει κανείς αυτό 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές. Δεν είμαι σίγουρη.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 Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε, συμφωνείτε μέχρι την 89 ε, όλες μαζί. Ωραία. 77 έως 89 όλες μαζί. Υπέρ. Α, τότε πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε και ξεχωριστά την κάθε λέει η πρόεδρος σε απάντηση παρατήρησης. 77 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, από 81 λοιπόν μέχρι 89 όλες μαζί. Ωραία. 89, 81 μάλλον, όχι 89, όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται 90, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 για την τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε λοιπόν την 92. Αρχίζει η ψήφος. Τέλος. Συφη 8 υπέρ 7 κατά εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά. Αποχές. Αν δεν σηκώνετε καθαρά το χεράκι σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας κάνουμε παλήθευση ηλεκτρονικά λοιπόν. 95. Δευτέρας Απορρίπτεται 7 υπέρ 9 κατά. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται 9-7. 97 τώρα. Υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι ήταν η ίδια ακριβώς πλειοψηφία όπως πριν 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση εν προκειμένου Τέλος. 9 κατά 7 υπέρ. Μου φαίνεται είναι πάντοτε η ίδια πλειοψηφία. 102 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι επόμενες τρεις δεν ψηφίζονται διότι είναι ταυτόσιμες με το κείμενο της εισηγήτρια. 112 λοιπόν υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται αυτή. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και αυτή τελική ψηφοφορία ονομαστική, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. 14 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Λοιπόν, μεγάλη πλειοψηφία ενεκρίθηκε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Η κυρία Μποσκόρ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια. Είμαι πολύ ευγνώμων για την υποστήριξή σας γιατί υπερψηφίσατε αυτή την γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί για μας ε, οι κοινότητες μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τύχουν υποστήριξης Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και τον βοηθό μου, ο οποίος συνέβαλε στην σύνταξη αυτής της έκθεσης των Φαμπιέν, γραμματεία και τους συνομιλητές καθώς και συμβούλους. Χαίρομαι για την ε, πολύ επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους. Η Πρόεδρος πάλι, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε και από την δική μου σκοπιά συγχαρητήρια για την δουλειά και της ηγήτριας και της κοιόδης ηγήτριας και βεβαίως και των μελών της γραμματείας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας προχωρήσουμε τώρα Η Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε στο θέμα 6 της ημερησίας διάταξης. Α, με συγχωρείτε, στο θέμα 5, 5 την παρουσίαση της μελέτης με τον τίτλο «Ψηφιακές ικανότητες στον 21ο αιώνα». πρέπει να, να προσέξω τώρα πάρα πολύ πώς θα ε, προφέρω το όνομα της κυρίας Γιουστίνα Βαϊκουτίτε Πασκαουσκέ. Ελπίζω να μην το ε, ε πρόφερα πολύ άσχημα το όνομά σας. Σας ε, καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Η κυρία Πασκαουσκέ προέρχεται από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Διοίκησης της Λιθουανίας. Θα δείτε λοιπόν ότι οι επόμενες τρεις ώρες Τη ε, συνάντησή μας είναι αφιερωμένες σε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πολύ υψηλά στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές δεξιότητες δηλαδή. Αρχίζω με την παρουσίαση τη σχετική μελέτη, δηλαδή ψηφιακές ικανότητες ή δεξιότητε στον 21ο αιώνα και μετά θα παρακαλέσω ε, την κυρία Μπενίνη και τον κύριο Δημητρόφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα οποία καλωσορίζω βεβαίως εδώ ε, να ε, εξηγήσουν την ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή οικονομία. Θα προχωρήσουμε μετά σε ένα γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων για να μπορέσουμε να περάσουμε αμέσως μετά στο υπαριθμό 6 της ημερήσιας διάταξης για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Πάντως, τώρα πρώτα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην εμπειρογνώμονά μας, κυρία Βαϊκουτιτέ Πασκαοσκέ. Δύσκολο, δύσκολο όνομα. Ομολογουμένω. Βέβαια είμαι σίγουροι ότι και ανάποδα θα σημαίνει το ίδιο. Δηλαδή και εσεί θα δυσκολεύεστε με την εκφορά των δικών μας ονομάτων. Έχετε λοιπόν 10 ε, λεπτά για να παρουσιάσετε την ε, μελέτη. Ορίστε, έχετε το λόγο κυρία Πασκάουσκε. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Πασκάουσκε. Σας ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή θα κάνω μια παρουσίαση για την ε, μελέτη μας για τις ψηφικές δεξιότητες του 21 ο αιώνα, μια γενική εικόνα της ε, έκθεσης. Μετά το σχέδιο δράσης για την ψηφική εκπαίδευση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2018, Στόχος μας ήταν ε, να δούμε την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, τις πολιτικές πρωτοβουλίες, να αξιολογήσουμε το προτινόμενη δράση, να εντοπίσουμε τα τυφλά σημεία και να παρέχουμε συστάσεις στην Επιτροπή. Οι πρώτε ε, προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στο σχέδιο δράση της Επιτροπή είναι η χαμηλή συνδεσιμότητα των σχολείων, τα μη επαρκή ε, προσόντα των ε, εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τα ψηφιακά μέσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ο λόγος είναι η έλλειψη αρχικής και κατά τη διάρκεια της εργασίας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς. Η αυτοαξιολόγηση θεωρήθηκε ως βασική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να υποστηρίξει και να αντιμετωπίσει αυτή την, ε, αυτό το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων. Αυτό το εργαλείο που ονομάζεται SELFI αφορά τα εκδευτικά, τους οργανισμούς για να αναπτύξουν ε, στρατηγικές αν ε, και εφόσον γνωρίζουν ποιες ε, είναι οι δυνάμεις τους ποιες είναι και ποιες οι δυναμίες τους. Η έκθεσή μας θεωρείται αυτή μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αλλά ότι χρειάζεται παράλληλα στήριξη μέσω διευθυντικών μεταρρυθμίσεων σε κρατικό επίπεδο και γι' αυτό η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα ε, στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν προγράμματα ε, εκπαιδευτικά για τους εκπαιδευτικούς. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που δεν εντόπισε η έκθεση είναι βεβαιότητα για τα θέματα των δικαιωμάτων διανοητικής διεκτησίας. Υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα ως προς το πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποιούν ε, τα υλικό, το ψηφιακό υλικό. Γι' αυτό θα χρειάζεται να έχουν μεγαλύτερη, περισσότερη εκπαίδευση, ειδικά μετά τη νέα οδηγία για το copyright που θα τεθεί σε ισχύ. Άλλες προκλήσεις είναι η έλλειψη ε, υπηρεσιών, ψηφικών υπηρεσιών που αφορούν ε, τους ε, μαθητές που βρίσκονται σε κινητικότητα. Υπό την έννοια ότι το σχέδιο δράσης προτείνει προτείνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου ώστε να επιστοποιούνται τα ψηφιακά προσόντα και να επικυρώνονται οι δεξιότητες. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και η συστάσεις μας είναι να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις για την ε, ε, διακυβέρνηση, την ενδεχόμενη διακυβέρνηση αυτού του προτύπου. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά ε, πρότυπα ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών, γιατί πολλοί οργανισμοί βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Άλλο θέμα που εντοπίσαμε είναι ότι θα χάσει ανταγωνισμό η αγορά εργασία αν το κρατικό σύστημα δεν μπορεί να ε, παράγει ε, και ε, ψηφιακέ δεξιότητε απλέ απλές και πιο προηγμένες. Μία από τις δράσεις που προτείνεται από το σχέδιο δράσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απο τι δρασεις που προτεινεται απο το σχεδιο δράση οτι θα πρεπει να υπαρχει μια πλατφορμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανώτατη εκπαίδευση και για ενισχυμένη συνεργασία. Δηλαδή, να υπάρχει μια πλατφόρμα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ανταλλάσσουν τις βαλίτσες πρακτικές και να ενθαρρύνουν την διεθνικοποίηση. Επίσης, προτείνεται η προσθέμενη αξία μιας τέτοιας πλατφόρμας συνεργασίας να συζητηθεί, ε, να εμπλέξει τα ενδιαφέρομενα μέρη πέρα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να μελετήσει συνέργειες με άλλες υπάρχουσες πληροφο... Ε, στρατηγικές που υπάρχουν. Ε, το χάρη με το Erasmus Plus ε, που ήδη στηρίζει την συνεργασία. Ένα άλλο θέμα που εντοπίσαμε στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση είναι ε, ο χαμηλός αλφαβητισμός, ψηφιακός αλφαβητισμός μεταξύ των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Επίσης, η διεύρυνση του ε, χάσματος μεταξύ των φίλων, όπου υπάρχει λιγότερη ενθάρρυνση για τα κορίτσια να ακολουθήσουν μια καριέρα στις θετικέ επιστήμες, τη τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, αλλά και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Το σχέδιο δράση προτείνει λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα να, να οργανωθούν ε, εργαστήρια για τα κορίτσια όπου θα τους παρέχονται θετικά πρότυπα και θα ενθαρρύνονται να επιδιώξουν σπουδέ στον κλάδο ICT και STEM στην καριέρα τους, να κάνουν μια καριέρα σε αυτό το τομέα. Όμως, ε, έβριμα της επιτροπή. Τη ε, έκθεση ε, ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική και ένα ξεκάθαρος οδικό χάρτη για το πώ θα ενισχύσουμε τη συνεργασία και πώ πώς θα ε, καταρτήσουμε δράσει ω προ αυτό το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για ένα στρατηγικό σχέδιο με σχεδιασμένε δράσει, και ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη χάρξη πολιτική, ε, πρωτοβουλίε ε, πολιτικών, χρηματοδότηση ώστε ε, αντιμετωπιστεί περαιτέρω αυτό το θέμα. Και τέλος, ε, τελικό σημείο στην ε, παρουσίασή μου είναι ε, κάτι άλλο που εντοπίστηκε και ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή ε, όσον αφορά τα δεδομένα για την ψυχική εκπαίδευση και το σχέδιο δράσης. Ε, προτείνει μια πληθώρα δράσεων να υπάρξει μια μελέτη αναφοράς ε, που θα αξιολογήσει την πρόοδο ε, στην εκπαίδευση σε σχέση με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, να προτεθεί ένα καινούριο μόντουλ στο πλαίσιο της ε, PISA και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι, είναι η ανάπτυξη των μεγάλων δεδομένων και των analytics. όλα αυτά θα μπορέσουν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες, πώς αυτά τα big data και τα learning analytics μπορούν να αξιοποιηθούν από τα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν η έκθεσή μας ε, θεωρείται θα ήταν αξιόλογο ότι εξίζει να αναλύσουμε, να, να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις του ε, Joint Research Center, του Κοινού Κέντρου Έρευνας, θα πρέπει να οριστούν προτεραιότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, να δημιουργηθούν πολυπληρωτικά προγράμματα, προγράμματα για Learning Analytics, να καθοριστεί ένα οδικό χάρτη χάρτης για το πώς θα αναπτυχθούν οι πρακτικές και οι δράσεις και τέλος ε, να βρεθούν οι συντονιστές και τα αρμόδια όργανα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σα σας ευχαριστώ και αν έχετε ερωτήσεις μπορούμε να τις ε, απαντήσουμε. Yeah, Ευχαριστώ πολύ για την ε, γρήγορη παρουσίαση. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν πολύ όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας. Τώρα περάσουμε στις... Ε, πρωτού περάσουμε στις ερωτήσεις, περάσουμε στους επόμενους εκπροσώπους της Επιτροπής. Ο λόγος Τώρα για να επεξηγήσουμε τι ε, πιστεύει η Επιτροπή για το σχέδιο δράσης, ε, για την ψηφιακή εκπαίδευση. Αναμένουμε με αγωνία να σας ακούσουμε. Έχουμε ρίξει μια ματιά ε, στο τι έχετε ετοιμάσει. Όμως είναι πάντα χρήσιμο και ευχάριστο να μας το εξηγούν αυτό οι εμπειρογνώμονες. Καλώς ήρθατε λοιπόν την κυρία ο, ο λόγος σε πρώτη φάση του κύριο Δημητρόφ. Από κοινού 10 λεπτά, εσείς ε, θα αποφασίσετε πώς θα μοιράσετε το χρόνο σας. Ο λόγος σας. Ευχαριστώ κύριε Κάμπραβερ. αξιότιμο μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια ακροασία Η Επιτροπή καλωσορίζει αυτή την πρωτοβουλία για να σας μιλήσουμε για το πρόγραμμα δράσης ψηφιακής εκπαίδευσης. Θα σας μιλήσουμε για το πρόγραμμα δράσης, το σκεπτικό πίσω από αυτό και ο, ο μιλητής δίπλα μου από την Γενική Διεύθυνση Connect θα λάβει επίσης το λόγο. Ε, θα αρχίσω λέγοντας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει ανταπόκριση με τα συστήματα της κοινωνίας και αυτό αφορά και την αγορά εργασίας. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία και έχει μεγάλη σημασία να συνοδεύουμε τους καταρτιζόμενους ή τους εκπαιδευόμενους. Δεν θα σας δώσω σωρία στατιστικών, θα σας δείξω ένα διάγραμμα. Βλέπουμε ε, πόσα smartphones ε, χρησιμοποιούν τα παιδιά μεταξύ 12 με 15. Βλέπετε ότι το 83% των παιδιών ε, έχουν ένα smartphone. Τώρα μπορεί να είμαστε πάνω από το 90%. Και γνωρίζετε αυτό τι σημαίνει 10 χρόνια πριν, ο αριθμός ήταν μηδενικός περίπου. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Πρόκειται για μία ε, μαζική σδυσδυτική ε, χρήση των ε, κινητών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μιλούν για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, με τον ε, ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν υπάρχει σωστή στάθμιση ή μόχλευση. Βλέπετε το ποσοστό όσων εργάζονται σε αυτό τον ε, τομέα. Έχουμε πάνω από 6% στη Φιλανδία και Σουηδία, αλλά υπάρχουν πολλές ε, χειρευόμενες θέσεις ε, πάνω από 500.000 ανάλογα με τις πηγές σας. Αυτό δεν είναι παραγωγικό για την Ευρώπη και για την καινοτομία καθώς και την ανάπτυξη. Αυτός ο μετασχηματισμός δίνει πολλές δυνατότητες έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι προσβάσιμη, τα μαθήματα να είναι προσπελάσιμα για όλους, ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν γνώσεις. Εν πάση περιπτώσει για την ψηφιακή εκπαίδευση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις τεχνολογίες. Θα πρέπει να πούμε ότι με αυτά τα στοιχεία φυσικά τα σχολεία δεν πρέπει να μείνουν πίσω, θα πρέπει να συμβαδίζουμε με το διαδίκτυο και τις μεγάλες καινοτομίε. Σήμερα βλέπουμε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στην κορονίδα των μελημάτων μας στο Γκέτεμπορκ η Επιτροπή μίλησε για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου μέχρι το 2025 και το πρόγραμμα δράσης ψηφιακής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε εκεί. Έχουμε τρεις προτεραιότητες. Καταρχήν και 11 δράσεις βεβαίως. Οι προτεραιότητες είναι να γίνει καλύτερη χρήση των ε, ψηφιακών τεχνολογιών για να υπάρχει καλύτερη διδασκαλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον υπεύθυνο αυτής της μελέτης. Θα πρέπει να πω επίσης ότι πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία πολλών γενικών διευθύνσεων μεταξύ Γενική Διεύθυνση Connect και Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, αλλά συμμετείχαν και άλλες γενικές διευθύνσεις. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον πρώτο πυλώνα. Θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση και την εκμάθευση. Επίσης θα πρέπει να μας βοηθήσει ιδιαίτερα για την εκπαίδευση και την εκμάθευση. Αλλά δεν γίνεται πολύ καλή χρήση. Αν και έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο, υπάρχουν όμως αποτυχίες γιατί δεν υπάρχει συνδεσιμότητα πάντα και φυσικά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και αρμοδιότητες, πώς να υπάρχει προσπελασιμότητα και φυσικά η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι θα λάβουμε υπόψη πολλές αρμοδιότητες. Πρόκειται για μια πρόκληση πολύ, με, πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Ένα στους πέντε νέους δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 90% των θέσεων εργασίας προαπαιτεί ψηφιακή εκπαίδευση. Και θα αυξάνεται το ποσοστό. Ξέρουμε ότι πολλές θέσεις εργασίας θα ε, προϋποθέτουν μία διαφορετική τάξη δεξιοτήτων και μόνο το 15% αφορά ε, γυναίκες, το οποίο δείχνει ότι επιδεινώνεται το πρόβλημα. Δυστυχώς, οι γυναίκες, τις γυναίκες εκπαιδευόμενες ή εργαζόμενες, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Τέλος, θα πρέπει να βοηθήσουμε στην βελτίωση της εκπαίδευσης και την καλύτερη ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψη. Αυτό γίνεται με δοκιμές, με πειραματισμούς, να δούμε τι δεν έχει κάνει στο παρελθόν και φυσικά να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για ορισμένε δράσεις πριν λάβει το λόγο η Φαμπρίτσια. Η πρωταρχική δράση είναι το SELFIE, το πρόγραμμα ε, SELFIE, που είναι ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία. Στις 25 Οκτωβρίου θα γίνει η επίσημη εκκίνηση, αν και ήδη έχει, έχουμε πειραματιστεί σε 10 χώρες για να δούμε κατά πόσο τα σχολεία είναι έτοιμα το σχολείο λοιπόν θα μπορούν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και αρμοδιότητες ολιστικά και να προωθήσουν προγράμματα δράσης. Αυτό θα το ξεκινήσουμε φέτος. Η δεύτερη δράση είναι η ανάγκη της, ε, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, και αυτό σημαίνει εργαστήρια για ε, τα κορίτσια στην ε, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή κορίτσια που θέλουν να ε, συμμετάσχουν στη συνέχεια στον επιχειρηματικό κόσμο. Και η τελική δράση αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση αυτής. Μιλάμε για την εφαρμογή ε, ε, μιας τεχνικής που λέγεται crawling, όπου βάζουμε στοιχεία στο σύστημα και να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να προγραμματίζονται, να προσχεδιάζονται τα μάστερ ή τα βασικά πτυχία. Τώρα θα δώσω το λόγο στη Φαμπρίτσια. Χωρίς μικρόφωνο, η ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί προσδίδεται μεγάλη σημασία στις ψηφιακές δεξιότητες. Έχει μεγάλη σημασία η δική σας οπτική γωνία και ματιά. Γενικά η DigiConnect θα εποπτεύσει το θέμα της συνδεσιμότητας και τις ε, δεξιότητες, ψηφιακές ε, δεξιότητες. Θα βρείτε λεπτομεριακές ε, πληροφορίες στον απογραφικό κατάλογο για να δείτε ποιος είναι ο βαθμός διείσδησης της συνδεσιμότητας. Αν δούμε το πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη δράση υπαριθμών 1 δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το ευρυζωνικό στα σχολεία, γιατί αν δεν υπάρχει θα είναι δύσκολο να συμμετέχουν οι φοιτητές, οι μαθητές και έχουμε ένα 80% των σχολείων που δεν έχουν αυτή τη συνδεσιμότητα. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει κατάσταση στα κράτη-μέλη. Καταρχήν να υπάρχει μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα έτσι ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να τύχουν χρηματοδότησης από το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω του ΣΕΦΤ συνδέοντας την Ευρώπη αλλά και μέσω του ΕΚΤ όπου γίνεται χρηματοδότηση των σχολείων και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα, επειδή υπάρχει ένα δίκτυο γραφείων ευρυζωνικότητας, θα μπορέσουμε να δούμε πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι διάβλοι. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα σχολεία μέσω της συνδεσιμότητας και στο επόμενο πολιετές το ΣΕΦ, το Συνδέοντας στην Ευρώπη, θα βοηθήσει για την χρήση των, ε, αυτής της δυνατότητας Gigabyte, τα οποία θα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των σχολείων. Τώρα, η δράση υπαριθμών 6 έχω ε, εγώ αυτή την κονκάρδα και θα ήθελα να βρείτε και εσείς γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ε, ε, του κώδικα που χρησιμοποιείται στα σχολεία. Είναι ένα ευρύ πλαίσιο από τις 6 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και στόχος είναι να, να έχουν πρόσβαση το 50% των σχολείων μέχρι το 2020. Να μπορέσουν να προωθήσουν τουλάχιστον μία ε, δράση σε αυτή την Code Week. Γιατί αυτό είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να μην είμαστε μόνο χρήστες ή καταναλωτές, να είμαστε και ε, δράστες. Ε, αυτή η εβδομάδα ισχύει για όλους, η Code Week, και θα δείτε στις διαφάνειες ότι υπάρχουν πολλά link και για τις επαγγελματικές πηγές και μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αυτών των δεδομένων μέσα στα πλαίσια της χαρτογράφησης για να μπορέσουμε να εποπτεύουμε επιγραμμικά. Θα ήθελα να δείτε πώς έχει μία συνεδρίαση των ε, επικεφαλής. Πρόκειται για μία σωρία ε, t-shirt διαφόρων χρωμάτων, όπου συμμετέχουν βεβαίως όλοι. Η τελευταία ε, δράση αφορά τις προκλήσεις της του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εδώ έχουμε ένα μακρύ κατάλογο Ποια είναι η ανταπόκριση, ποια είναι η απάντηση, ο τρόπος ε, ε ενδυνάμωσης και ε, μίας επικοινωνίας, μίας ε, εκπαίδευσης ενσυνειδητότητας. Θέλουμε οι νέοι, τα παιδιά, οι γονείς, οι δάσκαλοι να συμμετέχουν αυτή τη διαδικασία back to school, όπου τα παιδιά θα πρέπει να είναι αρκετά πειθαρχημένα, να έχουν μια υπεύθυνη θέση και στις 20 Νοεμβρίου θα έχουμε τους νικητές από αυτό το διαγωνισμό τον διαδικτυακό. Τώρα, ως προς τις γυναίκες στον ψηφιακό κόσμο είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Έχουμε μία στρατηγική και θα υπάρχει και μία ε, διαδικασία βαθμολόγησης των σχολείων. Ελπίζω τον επόμενο Οκτώβριο, την Πέμπτη θα γίνει παρουσίαση και ελπίζω να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα τον Οκτώβριο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και την κυρία και τον κύριο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και προχωρούμε τώρα σε ένα σύντομο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων και επειδή δεν είναι ιδιαίτερος πολύ άριθμα τα μέλη της Επιτροπής, ας μην είμαστε και τόσο τυπολάτρες, ώστε να πούμε μόνον οι σκιώδεις συγητές θα έχουν το δικαίωμα της λήψης λόγου. Όποιος έχει ερωτήσεις μπορεί και όποια να ζητήσει τον λόγο. Ενδεχομένως να δώσω πρώτα το λόγο στους σκιώδεις συγητές. Η εισηγήτρια της εκθέσεως πρωτοβουλίας δυστυχώς δεν έχει φτάσει ακόμη. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να έλθει μέσα στη διάρκεια του απογεύματος. Θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία την οποία λέμε εδώ ping-pong, δηλαδή θέτετε ερώτηση εφόσον επιθυμείτε και μας λέτε σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση συγκεκριμένα. Ακούτε την απάντηση και προχωρούμε. Και πρώτη έχει ζητήσει το λόγο κυρία Ροδρίγες. Κύριε Ροδρίγκε, έχετε το λόγο. Α πούμε για δύο λεπτά, αν μπορείτε. Θα σα τα πω στα πορτογαλικά. Παρακαλώ φορέστε ακουστικά. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και τις ε, δύο παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές. Τώρα, σε σχέση με την παρουσίαση της Ζουστίνα, εγώ ήμουν εισηγήτρια το 2015 για μία έκθεση πλαισίωσης των νέων κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης. Γιατί πολλές φορές τα κορίτσια δεν συμμετέχουν σε, αυτές τις, σε αυτά τα μαθήματα πληροφορικής. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βρίσκεται το καθεστώς των ποσοστώσεων, έτσι ώστε τα κορίτσια να συμμετέχουν στις νέες τεχνολογίες. Δυστυχώς σε αυτό το τομέα επικρατούν οι άντρες. Όμως στον τομέα της πληροφορικής, τουλάχιστον στην Πορτογαλία, η κατάσταση είναι πιο ισορροπημένη αλλά στον τομέα ε, της μηχανικής δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η, η ίδια ερώτηση αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απευθύνεται σε αυτήν. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές και ασχολήθηκα με τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, γιατί και εγώ προέρχομαι από μία από αυτές. Αυτά τα μαθήματα δεν φτάνουν στην, στις αίθουσες των απομακρυσμένων περιφερειών. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλές φορές ε, ε γίνονται μαθήματα, αλλά αναφέρονται μόνο γενικολογίες τα μαθήματα αυτά. Αυτό μου λένε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Άρα αυτές οι δράσεις φτάνουν και εντάσσονται σε παιδαγωγικές πρακτικές. Και πώς αντιμετωπίζετε την κοινότητα των ενηλίκων έτσι ώστε να διαθέτει περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η πρώτη σας ερώτηση απευθύνεται περισσότερο στην εμπειρογνώμονα που έχει συντάξει τη μελέτη, έτσι δεν είναι. Έχει το λόγο κυρία ε, Πασκάουσκε. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ήταν περισσότερο ένα σχόλιο για την ε, παρουσίαση εξετάσαμε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή δεξιότητα και το θέμα των κοριτσιών, των νεαρών ε, ε, κοριτσιών δηλαδή, ε, στην εκπαίδευση. Η έρευνα δείχνει ότι παρόλο που πολλά νεαρά κορίτσια παρακολουθούν τέτοια μαθήματα στην ε, πρωτογενή εκπαίδευση μετά εγκαταλείπουν την εκπαίδευση αυτή διότι δεν υπάρχουν ε, πρότυπα, δεν υπάρχουν δηλαδή μοντέλα ρόλοι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που οι γυναίκες να μπορέσουν να μιμηθούν ή να θέλουν να μιμηθούν. Επίσης υπάρχουν τα στερεότυπα ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι περισσότερο για τα αγόρια και τα κορίτσια ακολουθούν άλλες σπουδές. Μπορώ δηλαδή να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε ότι στις μικρές ηλικίε κορίτσια και αγόρια ε, ασχολούνται το ίδιο με coding και STEM κλπ. Μετά όμως εγκαταλείπουν σιγά σιγά τις σπουδές αυτές τα κορίτσια και διευρύνεται το κενό μεταξύ των δύο φίλων στο, στον χώρο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Δημητρόφ ή εσείς κύριε Μπενίνη, όπως επιθυμείτε. Κύριε Δημητρόφ, εσείς. Ευχαριστώ την κυρία Ροδρίγες για την ερώτησή της. Να αρχίσω με ένα γενικό σχόλιο για την ε, παρατήρηση που κάνατε για την γενική μας προσέγγιση και ρωτήσατε μετά πώς διασφαλίζουμε το monitoring και την παρακολούθηση του τι γίνεται μέσα στην ίδια την αίθουσα, τη σχολική αίθουσα. Εδώ βρισκόμαστε βέβαια πρώτα-πρώτα σε πλαίσιο επικουρικότητας. Ε, πρώτος εγώ το λέω αυτό και το τονίζω και νομίζω ότι πρέπει να το έχει κανείς πάντοτε υπόψη του όταν μιλεί για κατάρτιση και εκπαίδευση. Είναι πράγματι θέμα για το οποίο έχουμε ακούσει από πολλές χώρες μέλη στη διάρκεια των μηνών που πέρασαν από τον Ιανουάριο, για παράδειγμα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Bundesrat της Ομοσπονδιακής Γερμανίας έδεσε υπόψη μας ε, τη γνωμοδότησή του και ε, βεβαίως εμείς λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις υπόψη τις γνώμες αυτές. Η προσέγγιση μας είναι λίγο διαφορετική. Ο λόγος που προωθούμε το σχέδιο δράση είναι διότι συναπαρτίζεται από διάφορες δράσεις. Ορισμένε μπορεί να είναι πιο στενές. Ίσως να μην είναι τόσο σαφώ καθορισμένες με στο ίδιο το σχέδιο δράσεω. Στο μεταξύ έχουμε εκδώσει έναν αριθμό δελτίων που εξηγούν ε, το συγκεκριμένο περιεχόμενο της κάθε δράσης. Δεν είμαι σίγουρος εάν τα πανεπιστήμια έχουν όντως λάβει τα σχετικά έγγραφα όμω αυτά αποτελούν απόσπαστο μέρος του συνολικού πακέτου. Για το πώς θα φτάσουμε μέσα στη σχολική αίθουσα, πρώτα θα πρέπει να είμαστε σαφείς εάν όντω είναι δική μας υπόθεση να φτάσουμε στη σχολική αίθουσα. Αυτό ε, είναι πράγματι αλήθεια όταν πρόκειται για ανταλλαγή ευέλικτων ε, πρακτικών, όπως με το ε, σύστημα selfie, όπου είχαμε ένα καλό ε, σκορ πέρσι, δηλαδή 60.000 μαθητές και διδάσκοντες και γι' αυτό έχουμε βάλει ως στόχο το 1 εκατομμύριο στο τέλος πλέον του χρονικού πλαισίου του σχεδίου δράσεως. Υπάρχουν λοιπόν εξειδικευμένες δράσεις που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε μέσα στη σχολική αίθουσα, οι οποίες ποτέ δεν μπορούν να λύσουν ολόκληρο το πρόβλημα. Πρόκειται για μια σταγόνα, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια που ελπίζουμε ότι θα ε, επηρεάσουν για την ε, διδασκαλία των ενηλίκων. Τέτοια σχόλια έχουμε ακούσει και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Λάβαμε εν συνείδητη απόφαση να περιοριστούμε στην τυπική διδασκαλία, αλλά όχι την διαβίου κατάρτιση. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όμως, λόγω του χρονικού πλαισίου του σχεδίου δράσεω, το οποίο αναφέρεται σε δράσει μέχρι το 2020, και δεν προκαταλαμβάνει το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μην στοχεύσουμε στη γενικότερη εικόνα, γιατί ε, χρειάζεται την προσοχή μα. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε όμω σύντομε και σύντομοι, διότι αλλιώ ε, θα ε, σημειωθεί καθυστέρηση. Ορίστε, κύριε Μπενίνη. Να επαναλάβω ότι Υπάρχει αυτή η στρατηγική για τι γυναίκε στο ψυχικό τομέα και είναι κάτι που το λαμβάνει πολύ σοβαρή υπόψη η επίτροπο μου που είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε τρει άξονε. Ο ένα είναι να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα μεταξύ φίλων. Πολλά κορίτσια έρχονται σε αυτόν τον τομέα τη εκπαίδευση αλλά δεν τον ολοκληρώνουν. Γι' αυτό εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα και θέλουμε παράλληλα να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να μάθουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό. Γι' αυτό θα απονείμουμε και κάποια βραβεία το 2019 και υπάρχει και μια άλλη πτυχή που ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και εκεί υπάρχει ένα δίκτυο γυναικών που είναι γυναίκες επιχειρηματίες και παράλληλα ξεκινάμε στέλνοντας μια πρόσκληση σε CEOs ώστε να προχωρήσουμε σε μια διακήρυξη που θα προωθήσει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες στον κλάδο αυτό. Είναι δράσεις που από κοινού θα μπορέσουν να επιφέρουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μαλίνο. Προσπαθήστε και εσείς να περιστείτε στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρα σύμπτωση ε, ότι μόλις ήρθαμε από το Silicon Valley και είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι θα ήμασταν. Είναι πραγματικά επιλεκτικό γιατί έχουμε το, τις ίδιες ε, παρουσιάσεις στα κεντρικά της Apple. Έχουν ε, λίγο διαφορετική ορολογία. Μιλάνε για developers, για digital developers. Αλλά μιλούσαν για το τι κάνουν στον τομέα της εκπαίδευσης και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο προχωρημένη οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως αναρωτιέμαι, παρουσιάζονται δύο ποσοστά, 40% του εργατικού δυναμικού θα χρειαστεί δεξιότητες, τα 40% των μελλοντικών επαγγελμάτων θα συνδέονται με ψηφιακή δεξιότητε, αλλά δεν ξέρουμε ποιε θα είναι αυτές οι θέσει εργασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εκεί που μας έγινε η παρουσίαση, δεν, παρουσίασα, δεν παρατήρησα τη αναλογία μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στο πανεπιστήμιο. Πώς το κάνουν αυτό, έχουν ποσοστώσεις, έχουν καλύτερα τεστ, ώστε να είναι πιο δίκαια. Δεν είδα όμως κάτι περίεργο. Τώρα, ε, αυτό που θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα, γνωρίζουμε όλοι, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πέρα από τις προσπάθειες μας και παράλληλα με αυτές, υπάρχει μια άλλη διαδικασία που λαμβάνει χώρα και που ηγείται ε, από τις επιχειρήσεις τον ειδικό τομέα. Είμαστε πίσω ως προς την παραγωγή, την απαραίτητη ποσότητα ανθρώπων που θα χρειαστούν δεν αναμένουν πλέον τίποτα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Λένε απλά 10% θα είναι από τις επίσημες δομές, τις εκπαιδευτικές. Δικιά μας είναι αυτή η πρωτοβουλία. Και παράλληλα δημιουργούν τις δικές τους δομές εκπαίδευσης. Και αν δούμε τις δομές αυτές, Δεν θέλω να πω κάτι κόλλη, είναι παράνομε. Αλλά είναι όμω παράλληλα πολύ πιο χρήσιμε και πολύ καλύτερε από οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε εμεί. Αυτό είναι το δικό μου το παράδοξο. Είναι κάτι με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε. Πρόεδρο, ποιο θα ήθελε να σχολιάσει το παράδοξο του κ. Μαλινόφ. Η κυρία Μπενίνη πρώτη. Κοιτάξτε, περιγράφετε την πραγματικότητα όπως είναι πραγματικά. Εμείς αναμένουμε από την επίσημη εκπαίδευση στο εθνικό επίπεδο, στο περιφερειακό επίπεδο. Βεβαίω θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό είναι εντολή των χωρών μελών μας και δική μας. Αλλά οι ψηφιακές δεξιότητες και οι εργαζόμενοι σε ψηφιακές δεξιότητες είναι ζήτημα που προωθούν τις δεξιότητες αυτές, δηλαδή και την απόκτησή τους, οι ε, ιδιωτικές εταιρείε από μόνε του. Αν μιλείτε για το αμερικανικό παράδειγμα, το πρόβλημα συχνά είναι ότι από τη στιγμή που εκπαιδεύεται ένα εργαζόμενο, αντιμετωπίζει ρήτρε που του απαγορεύουν ή της απαγορεύουν να μετακινηθεί σε άλλη δουλειά από εκεί όπου του έχει χορηγηθεί η τις απαγορευουν να μετακινηθει σε αλλη δουλεια απο εκει οπου του εχει χορηγηθει η εκπαιδευση Το εξετάζουμε αυτό. Εξετάζουμε και τη μεταφορά ε, γνώσης ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στον δικό μας τομέα. Και αυτό είναι συμπυκνωμένο με το νόημα της ε, δράσης μας που ε, βασίζεται στην ανάπτυξη high-end technology, HSPC, cyber security και βεβαίως υπάρχει και μια πτυχή που αναφέρεται στις δεξιότητες. Εκεί όμως η διάδραση και η ε, σύγκριση στην προσπάθεια είναι μεταξύ χωρών μελών, βιομηχανίας, ειδικών και βέβαια για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Ε, έχει ενστερνιστεί την ανάγκη να συνδέσει τι βιομηχανικέ εξελίξει, τι οικονομικέ εξελίξει με την στήριξη τη απόκτηση δεξιοτήτων. Αυτά τα έχει λάβει πόση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα έχει ενστερνιστεί, όπω είπα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ Πέτρα και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μαλινόφ, γιατί και εγώ πήγα μαζί με την αντιπροσωπή αυτή στην Silicon Valley και βρέθηκα πραγματικά σε αυτό το πολύ προηγμένο μέρος ε, του ε, ε, ψηφιακού καπιταλισμού. Και είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στο τι συζητούμε εδώ και πώς τα συζητούμε. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά. Τουλάχιστον. Γι' αυτό θα ήθελα, συμφωνώ μαζί σου ότι χρειαζόμαστε ψηφιακή εκπαίδευση, σχέδιο πανευρωπαϊκή συνειδητοποίηση, ζητήματα media literacy, ασφάλεια, κυβερνοασφάλειας κλπ. κλπ. Και χρειάζεται να ενισχυθούν οι δεξιότητε. Ακούγοντα σα όμως το mindset, η, διάθεση, η προετοιμασία για να δράσουμε, πώς να πω, δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση που είδαμε με τα μάτια μας την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, έχω και συγκεκριμένες ερωτήσει. Μιλήσατε για το MOOCs, Massive Online Courses ε, τα συζητούσαμε αυτά 10 χρόνια και το feedback που λαμβάνω εγώ είναι ότι χρειάζεται κανείς πάντοτε ένα συνδυασμό reskilling και upskilling με ιδιαίτερε ικανότητε για του ε, διδασκόμενου, αλλά χρειάζεται κανεί απαραίτητα και πολύ καλού διδάσκοντε. Διότι ε, πάνε να ε, φτιάξουν αναλογικέ σχέσει με ψηφιακά εργαλεία. Τελικώ όμως μην λησμονείτε ότι χρειάζεται πραγματικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία. Ε, δεύτερη ερώτηση. Η ανάγκη να επιταχύνουμε. Είναι δεδομένη. Όταν βλέπει κανείς πώς πήγαμε και είδαμε Apple, Facebook, Google, Airbnb, ε, Netflix και τα πανεπιστήμια, Stanford και Berkeley και μη κυβερνητικέ οργανώσει που ξέφυγαν ε, ε, ε, από του μεγάλου αυτού γίγαντε, γιατί είπαν ότι αυτά που κάνουν είναι πολύ επικίνδυνα. Βεβαίω πρόκειται για πανεπιστήμια elite όπω Stanford και αυτά. Η διασύνδεση του όμω με τι εταιρείε είναι πάρα πολύ στενή. Έχουν δηλαδή πάρα πολύ διαφορετική πολιτική και επιχειρηματική νοοτροπία έχουν κάτι που ε, δεν έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή μαθαίνουν από τις αποτυχίες τους, μια και δυο, και όλα αυτά με risk skill, up skill, ε, ε, μαθητές, φοιτητές κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε, διότι τα επιβάλλει ο ανταγωνισμός. Από την άλλη μεριά, όταν μιλούμε για ψηφιακή στρατηγική, θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Άρχισα μόλις να διαβάζω ε, το νέο βιβλίο του Ισραηλινού καθηγητού Χαράρη που λέει 29 ερωτήσεις για τον 21ο αιώνα και αυτή η βιοψηφιακή ε, επανάσταση τι θα γίνει, πού θα πάει, ε, είναι σαφή τα πράγματα αυτά. Αυτό λέει ο Πανεπιστημιακό Καθηγητής. Όλα αυτά θα είναι δεδομένα, αλλά χρειαζόμαστε ανθρώπου, ανθρώπινα όντα τα οποία θα αποφασίζουν τι θα γίνουν με αυτά και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να κρίνουν για τη χρήση των τεράστιων αυτών ποσοτήτων δεδομένων. Και αυτό το πρόβλημα εσείς δεν το αναφέρατε καν. Και αν μιλείτε για στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπω πρέπει να διευρυνθεί η εικόνα που έχουμε του θέματο. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Αλλά παρακαλώ σύντομα κύριε Δημητρόφ. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε την Apple, το Netflix κτλ. Ναι, φυσικά είναι δύσκολο να συγκριθούμε με αυτές τις εταιρείε που είναι στην κορυφή και παραμένουν στην κορυφή. Θεωρώ ότι τα κριτήρια αναφοράς είναι πολύ μεγαλύτερα και Μελετάμε και την πτυχή της συμπερίληψης ώστε να είναι προσβάσιμος ο κλάδος σε όλους. Φυσικά και είναι πολύ πιο προηγμένη σε σχέση με εμάς. Συμφωνώ με αυτή την αξιολόγηση. Σε αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ μετά από πέντε χρόνια από την πλευρά της Επιτροπής δεν είχαμε πολιτική πρωτοβουλία ε, σε αυτόν τον κλάδο το 2013. Έχουμε όμως μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση το κάναμε το 2018 ε, μέσω του κολεγίου. Δεν είναι καλύτερη, ε, καλύτερο, το καλύτερο timing, όμως είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ε, σπέρνουμε τους πόρους για το μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν που το δείξατε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι στην επόμενη Επιτροπή θα ληφθεί πολύ πιο σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα όσον αφορά κυρίως την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό τους δασκάλου. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ε, παραδείγματα για το πώς βάζουμε στο, ε, στην πρώτη γραμμή τους ε, ε δασκάλους. Υπάρχει πλατφόρμα με παραπάνω από 400.000 δασκάλους που συνεργάζονται και ε, χρησιμοποιούν τις ε, πλατφόρμες αυτές τις ψηφιακές εδώ και 10 χρόνια και οι αριθμοί φυσικά αυξάνονται. Είναι αρκετά γρήγορα. Υπάρχει όμως αυτή η εξέλιξη, γίνεται και θέλουμε να προοδεύσουμε. Όσον αφορά την συνεργασία με το Στάνφορντ κτλ. Γνωστά παραδείγματα, θα ήθελα να πω ότι έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα στην Ευρώπη και ένα από αυτά είναι είναι η Ευρωπαϊκή για την καινοτομία και την τεχνολογία που φέρνει τις επιχειρήσεις ε, πολύ κοντά σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή συνεργασία. Χρειαζόμαστε περισσότεροι. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Όχι όσο θέλαμε ενδεχομένως. Κυρία Μπενίνη, παρακαλώ. Να προσθέσω λοιπόν, ε, αν δούμε πέρα από το σχέδιο δράση για την εκπαίδευση, υπάρχουν όλες αυτές οι ερωτήσει που θίξατε και εξετάζονται στην DigiConnect μαζί με καθηγητές, εμπειρογνώμονε, επιχειρηματίε και σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου ασχολούνται με τον αντίκτυπο που θα έχει η ψηφιοποίηση στο μέλλον και αυτό είναι κάτι που θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του επόμενου έτους και ένα άλλο, μια ομάδα εργασίας για τις επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρετε είναι και δικές μας ανησυχίες. Δεν λέω ότι έχουμε τις απαντήσεις, όμως είναι κάτι το οποίο διερευνούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στην κυρία Πασκάουσκε. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Κύριε Πασκάουσκε, δεν έχω κάποιο γενικό σχόλιο, αλλά σύμφωνα όσα είπατε, ναι, υπάρχει ανάγκη για περισσότερε δεξιότητε και πιο προηγμένε. Και αυτό που είδαμε στην έρευνά μα είναι ότι η ψηφιακή εκπαίδευση και το σχετικό σχέδιο δράση μελετάει τα προ... τις προηγούμενες δεξιότητες και πώς μπορούμε αυτά να τα παρέχουμε στον πληθυσμό και από την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά ως προς ερευνητικό, την ερευνητική προσέγγιση πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τους πολίτες ε, στον τομέα αυτό να παρέχουμε ε, κατάρτιση για δεξιότητες από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση. Θεωρώ ότι η έμφαση που δίνεται στην ευρυζωνικότητα είναι πολύ σημαντική. Ειδικά σε εκλογικέ περιφέρειες όπως είναι η δικιά μου, που είναι αγροτικές περιοχές και ε, μας έχουν υποσχεθεί τοπικές αρχές ότι θα το διορθώσουν το θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως ε, ακόμα σημεία όπου δεν υπάρχει ε, ταχεία πρόσβαση. Αυτό είναι και ο ρόλος φυσικά των βιβλιοθηκών και αυτό που αναφέρεται για τις γυναίκες. Θέλω όμως να θίξω ένα άλλο θέμα της πρόσβασης όσον αφορά τις γλώσσες γιατί ήμουν πρόσφατα συζητητρία σε μια έκθεση που εγκρίθηκε στην τελευταία ολομέλεια που κάνει λόγο για την ψηφιακή εποχή και την τεχνολογία των, στον γλωσσολογικό τομέα. Είναι μικρός αριθμός των γλωσσών που κυριαρχούν ε, στις online υπηρεσίες και στο ίντερνετ και σε επίπεδο ε, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το να χρησιμοποιούμε μία γλώσσα που τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα και αν υπάρχουν τεχνολογίες για να τις χρησιμοποιήσουν, τότε αυτό δεν αρκεί. Γιατί η γλώσσα είναι λάθος, γιατί δεν μιλούν όλοι αγγλικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί Μπορεί να έχουμε στην Google στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μέλλον. Αυτό θεωρώ πως είναι κάτι που θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή και ειδικά αυτή την πτυχή των ψηφιακών δεξιοτήτων, γιατί είναι κάτι που θα μπορούσε να ε, δώσει όθηση στην οικονομία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα δώσει όθηση και στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημητρόφ ο Επίτροπο μου λαμβάνει υπόψη πολύ σοβαρά αυτή την πτυχή και το εργαλείο για το οποίο, στο οποίο αναφερθήκα το selfie θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, θα είναι μεταφρασμένο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Άρα θεωρούμε σημαντικό όταν υπάρχουν τέτοιου είδου εργαλεία για εκπαιδευτικού οργανισμούς σε όλες τι δυνατέ γλώσσε. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια Κώστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσδώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και υπάρχουν ε, τρία βασικά ερωτήματα. Και εγώ συμμετείχα στην ε, αποστολή στο Silicon Valley στις ΗΠΑ θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και από πλευράς λογισμικού στα πλαίσια αυτής της ψηφιακής επανάστασης που γνωρίζουμε ε, τα δέκα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτό που μας ε, απασχολεί είναι και οι κανόνες που θα ισχύουν για το διαδίκτυο, καθώς και για τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Ξέρουμε ότι φυσικά θα πρέπει να δημιουργηθούν οι δεξιότητες και η γενικότερη εκπαίδευση επενδύοντας στους ε, δασκάλους, το διδακτικό προσωπικό γενικότερα, αλλά ξεφεύγουμε λιγάκι από το αρχικό σκεπτικό που ήταν όλα για την τεχνολογία και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Μην ξεχνάμε φυσικά και το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει. Ως προς τα κορίτσια μέσα στα πλαίσια αυτής της ενδυνάμωσης. Υπάρχει αυτό το χάσμα και στην ε, επόμενη γενιά, στη νεότερη γενιά. Το άλλο θέμα είναι της ε, κωδικοποίησης ε, και της πρόσβασης στην πληροφορική. Έχουμε επικεντρωθεί στην κωδικοποίηση πρωτίστως, εντάξει, το selfie και όλα τα άλλα μέσα. Αλλά αν θέλουμε να υπάρχει κριτική σκέψη και συμπληρωματικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να ερμηνεύουμε ένα περιβάλλον, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να προτρέχουμε και όχι μόνο να προσαρμοζόμαστε εκ των υστέρων. Νομίζω ότι αργούμε κάπως, αλλά προσπαθούμε να προσδώσουμε σημασία και στα ψηφιακά μέσα, σε αυτή την ψηφιακή εργαλειοθήκη, έτσι ώστε η Επιτροπή να τα λάβει υπόψη και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποιο σημείο βρισκόσαστε, ποια είναι τα νέα μέσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρόφ, κύριε Μπενίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα για τα σχόλια. Σχετικά με το coding, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η δεξιότητα. Θέλω να προσθέσω μια πτυχή ότι είναι μια δεξιότητα που συνεχώς αλλάζει. Κάνουμε πολλές φορές λόγο για υπολογιστική σκέψη, computational thinking. Είναι μια πιο ευρία έννοια που έχει να κάνει με ε, λογική και ουσιαστικά τις ρίζες του coding. Ε, κάνουμε από κοινού έρευνες μαζί με το GRC να δούμε πώς μπορούν να πλαισιωθούν μελλοντικά σαν έννοια οι ψηφιακές δεξιότητες όσον αφορά το χάσμα κάνατε λόγο για το χάσμα των γενεών και φυσικά για τις ε, μειονεκτούσες ομάδες υπάρχει και μία άλλη πτυχή όσον αφορά το χάσμα ε, ως προς αυτούς που πραγματικά έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουν με την τεχνολογία. Ίσως ακούσατε στην επισκεψή στη Silicon Valley ότι για κάποιες αυτές τις εταιρείε ο καταναλωτής είναι το προϊόν. Και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβαίνει, ότι θα έχουμε τη γνώση και την ευαισθητοποίηση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, γιατί τον περισσότερο χρόνο τον περνάνε σε συσκευές και να προσέχουν τι κοινοποιούν, γιατί πολλοί επωφελούνται από αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μάλλον θα σταματήσω εδώ ε, με τα σχόλια. Κυρία Μπενίνη, αυτό που περιγράφεται είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, το coding, ο προγραμματισμός, είναι κάτι που εξελίσσεται. Πρέπει να ε, αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να μην τον αντιμετωπίσουμε σε μια άγνωστη, ε, άγνωστη έννοια. Σε κάποιους τομείς δεν υπάρχει το coding. Θα το αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά προσπαθούμε πάντα να ακολουθούμε τις τελευταίες τεχνολογίες, να μην μένουμε πίσω. Και έχοντας αυτό υπόψη, ο ρόλος των δημόσιων φορέων εκπαίδευσης Υπουργείων και των δράσεων αποτελεί ρόλο κλειδί. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφήσουμε να σταθεί εμπόδιο στην εξέλιξη της ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρώπης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, θα πω πλέον το όνομά σας, Γιουστίνα. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα έχει να κάνει πιο πολύ με την χάραξη πολιτικής. Εγώ αναφέρθηκα μονάχα στο τι είδαμε εμείς στην ερευνά μας στο σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης προβλέπει, ε, κάνει προστατικές προβλέψεις για το μέλλον αυτό το κομμάτι του σχέδιου δράση είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει να εξελιχθεί λίγο περισσότερο προ το πώς θα πετύχει αυτή την πρόγνωση και πώς θα είναι πιο εστιασμένο σε συγκεκριμένες στρατηγικέ για να παρέχει στον ευρωπαϊκό πληθυσμό τις απαραίτητες φυσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για το μέλλον, που θα χρειαστούν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια θετική κίνηση αλλά φυσικά χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί, όχι στο ε, κοντινό μέλλον, αλλά σε 5 ή 10 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία, ε, ευχαριστούμε πολύ ο στην κυρία Μπίλντ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τους ε, παρεμβαίνοντες. Το πρόγραμμα ψηφιακής δράσης λαμβάνει υπόψη τα παιδαγωγικά ε, λόμπι που ισχύουν ε, μέσα στα πλαίσια ενός σύρμου που ισχύει στη ΣΥΠΑ και δεν παρευρέθηκα στο Silicon Valley. Φυσικά θα πρέπει να, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες πληροφορικής ε, και φυσικά χρειαζόμαστε και χειρουργούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διδάσκουμε ιατρική από το δημοτικό. Στην ε, Φλόριντα είχε προταθεί οι μαθητές να μη συμμετέχουν στο πρόγραμμα ξένων γλωσσών τη στιγμή που ασχολούνται με την πληροφορική. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλος φόρτος προς τους μαθητές. Ας δούμε τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά σχολεία. Ποιες είναι οι προτάσεις σας έτσι ώστε να υπάρχει προγραμματισμός και ποια μαθήματα θα διακοπούν. Δεν φοβόσαστε ότι αυτή η διδασκαλία είναι απαρχαιωμένη τη στιγμή που οι μαθητές που την ε, παρακολούθησαν θα πρέπει να μπουν σε μια αγορά εργασίας όπου επικρατεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο ε, Κύριος Δημητρόφ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Λοιπόν, ρωτήσατε αν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα θα ζημιωθούν ε. εξαιτίας του coding. Δεν είναι αυτό που παρατηρούμε στην ε, μελέτη μας. Αντιθέτως, ε, οι καλά ε, ενσωματωμένοι και ολοκληρωμένοι ε, μαθήματα πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν. Η μελέτη των ξένων γλωσσών είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Γνωρίζετε τις διάφορες εφαρμογές και εργαλεία τα οποία είναι δωρεάν και προσβάσιμα και που είναι πολύ γρήγορα και βοηθούν στη μελέτη των γλωσσών. Δεν γνωρίζω το, το παράδειγμα της Φλόριντα που αναφέρατε, αλλά δεν σημαίνει ότι ε, θα αποβούν όλα αυτά εις βάρος άλλων μαθημάτων. Και δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά τη δεύτερη ερώτησή σας. Αν την σημείωσα, ίσως θα θέλετε να την επαναλάβατε ή... Την επαναλάβετε. Παρακαλώ. Δεν φοβόσαστε ότι αυτή η διδασκαλία έχει γίνει απαρχαιωμένη τη στιγμή που οι μαθητές θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας με βάση την τάχιστη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, είναι κάτι που μας ανησυχεί και υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό όντως συμβαίνει. Δεν θεωρώ που μπορούμε να κάνουμε εμεί από μόνοι μα, αλλά αυτό θα πρέπει να κάνουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτό που θα έρθει. Υπάρχουν στατιστικέ και δεδομένα για αυτόν τον κίνδυνο. Και μια μελέτη του περασμένου έτους υπολογίζει το 30% των διάφορων δεξιτήτων για επαγγέλματα σε 10 χρόνια θα είναι εντελώ καινούρια, άρα δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση το θέμα είναι να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο γιατί ε, ο μετασχηματισμό αυτό είναι ραγδαίο και πολύ ισχυρό. Άρα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε πάρα να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση και από μένα ή μάλλον παρατήρηση που θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συζητήσουμε και στο δεύτερο γύρο. Και το ερώτημά μου είναι ότι κάνετε λόγο για έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα του ICT, όπου μας λείπει εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν αποδείξεις αν αυτό το εργατικό δυναμικό μπορούμε να το βρούμε στον ακαδημαϊκό τομέα ή στο μη ακαδημαϊκό τομέα. Υπάρχουν ε, ε, αποδείξεις ότι στη Γερμανία ότι η έλλειψη που υπάρχει δεν ε, θα καλυφθεί από τον, τον ακαδημαϊκό τομέα. Και επίσης, όσον αφορά τη μελλοντική επαγγελματική κατάρτιση, τι σημαίνει αυτό και ε, ψηφιακές δεξιότητες για μένα είναι κάτι παραπάνω από το να μπορεί κανείς να κάνει προγραμματισμό, ε, να μπορεί να γράψει κάποιο ένα αλγόριθμο, αλλά να ξέρει και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό δεν είναι από μόνο του digital skills. Έχει να κάνει και με τον μύτο τεχνολογικό τομέα. Θα ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί. Δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνο μου. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από, αυτού, πίσω από αυτό ποια είναι τα συμφέροντα και να μάθω να μπορώ να διαχωρίζω το από το λάθος. Αυτή είναι μια εστίαση που θα πρέπει να έχουμε στην εκπαίδευση για τις ψηφιακές ε, δεξιότητες. Και όχι μόνο τον τεχνικό, τον καθαρά τεχνικό τομέα της εκπαίδευσης, του προγραμματισμού αλλά να υπάρχει μέσα και η έννοια της κριτικής σκέψης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τελευταίο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα για το χάσμα και πού βρίσκεται αυτό για τους έχοντες ψηλά προσόντα. Το χάσμα δεν υπάρχει, υπάρχει στο μήνα καθημερικό τομέα. Συγκλίνουν οι έρευνε στη Γερμανία και στι άλλε χώρες. Στον ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν δεξιότητες για open access που θα στηρίξουν το σχέδιο δράση. αλλά όσα, όταν μιλάμε για τη γενική εικόνα, το μεγάλο χάσμα βρίσκεται ε, στον επαγγελματικό κλάδο, στις startups, ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις και σίγουρα όχι στον ακαδημαϊκό κλάδο. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση και είναι κάτι που θα πρέπει να το καλύψουμε ε, και το καλύπτουμε στο σχέδιο δράσης. Θα μπορούσαμε όμως να το εξελίξουμε και παραπάνω. Σαν αφορά το δεύτερο ερώτημα, συμφωνώ με την αξιολόγησή σας ότι αφορά περισσότερα από τις προγραμματιστικές δεξιότητες και ένα από τα εργαλεία που έχουμε προβλέψει είναι το πλαίσιο ψηφιακών δεξιότητων που αφορά όλους τους πολίτες και το οποίο αφορά τα, διαφορά, τα διαφορετικά τμήματα του τι είναι ψηφιακές δεξιότητες, το να μπορούμε να εφαρμόσουμε κανόνες λογικής, και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το ε, για το programming και μεταγνωστικές ε, ικανότητες για, επίσης ε, για το τι κοινοποιούμε και πόσο μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό αλφαβητισμό είναι ένας κινούμενος στόχος ουσιαστικά αλλά με το πλαίσιο το οποίο ε, έχουμε δημιουργήσει μαζί με το GRC και πώς ακούμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο που παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση ε, σε σχέση με αυτές τις δεξιότητες. Το συντομότερο δυνατό παρακαλώ. η μεταμόρφωση τη οικονομία μα έχει μεγάλο δικτυπό στι ε, δεξιότητε αυτέ. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι τομεί που θα καλύπτονται, αλλά είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελκύσουν περισσότερο κόσμο που θα εργαστούν ε, στον κλάδο αυτό και να μπορέσουν να εξυπηρήσουν όλα αυτά τα ψηφιακά έργα. Έχουμε μια πρωτοβουλία που είναι ένα είδο και έχει αυτό το στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχουν ε, ε, θέσεις πρακτικής για τους ε, φοιτητέ, για τους ελκύσει, τους ελκύσουμε και όσον αφορά αυτό που είπατε για τον αλγόριθμο, φυσικά η διαφάνεια των αλγοριθμών είναι κάτι που το μελετάμε και το ερευνάμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. κυρία Πασκάουσκε, για το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και όπως και είπαν οι συνάδελφοι της Επιτροπής, οι ψηφιακές δεξιότητες δεν σημαίνουν πλέον ότι γνωρίζει κανείς πώς να κωδικοποιεί και να εργάζεται με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ίδιο σημαίνει, συμβαίνει και για την εκπαίδευση όταν μιλούμε για σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να την εξετάσουμε από μια ευρύτερη σκοπιά, από την ψηφιακή οικονομία δηλαδή, από την αυξανόμενη ε, σημασία των μεγάλων ε, εταιριών που ασχολούνται με την ψηφιακή οικονομία. Και το σχέδιο δράσης παρουσιάζει τις ε, ψηφιακές δεξιότητες μέσα από ένα πλήθος οπτικών, όχι μόνο των τεχνικών, αλλά χρειάζεται μια ευρύτερη προοπτική. Βεβαίω και χρειάζονται περαιτέρω βήματα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται η ε, ψηφιακή εκπαίδευση και όχι μονάχα από τη σκοπιά των ιδρυμάτων που ασχολούνται με αυτήν, γιατί τώρα έχουμε μπει σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων μερών και φορέων που ασχολούνται με την ψηφιακή εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ για το πρώτο αυτό και πολύ ενδιαφέρον μέρος του σημερινού απογεύματος. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητρόφ, την κυρία Μπενίνη, την κυρία Πασκάουσκε. Πολύ ευχαριστώ να παραμείνετε εδώ. Όμως θα θέλαμε να αλλάξετε θέσεις, να έρθει εδώ στα έδρανα του Προεδρείου το δεύτερο πάνελ, από το οποίο αναμένουμε να ε, μας αναπτύξει και άλλες ενδιαφέρουσες ε, οπτικές γωνίες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Βεβαίως, ε, ξαναλέω, μπορείτε να παραμείνετε και να παρακολουθήσετε την συζήτηση και θα παρακαλέσω να προσέλθουν ο κύριος Τουράντο, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, την κυρία Ιλώνα Κίσ, επικεφαλής προγράμματος δημοσίων βιβλιοθηκών 2020 του Ιδρύματος ε, Γράφω και Διαβάζω εδώ στις Βρυξέλλες και τον κύριο Δομήνικο Κόρτα που είναι εισηγητής από την Επιτροπή Περιφερειών ε, Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο δηλαδή ε, για θέματα ψηφιακής παιδείας. Ελπίζω ότι τα πρόσωπα αυτά είναι όντως παρόντα στην αίθουσα και ότι θα έλθουν να καθίσουν εδώ κοντά μας. ohne große Umschweife. Χωρίς καθυστέρηση, να περάσουμε παρακάτω. Να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Ντουράντο, όπως είπαμε, είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. Και για τους αδέλφους που δεν το έχουν κοιτάξει, έχουμε στις Βρυξέλλες ένα μια ψηφιακή τάξη ε, που χτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Αξίζει πραγματικά μια φορά να το επισκεφτείτε, να δείτε πώς θα μπορούσε να είναι το μελλοντικό σχολείο. Οι σχολικές επισκέψεις ε, μας δείχνουν ότι το σχολείο είναι το ίδιο. Όπως και πριν από πόσα χρόνια που τελείωσα εγώ το σχολείο, όμως χαιρόμαστε που είστε εδώ κύριε Ντουράντο, για να μας πείτε πώς θα είναι η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, πώς θα πρέπει να είναι. Κύριε Ντουράντο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε για να μοιραστούμε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες και πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Θα ήθελα καταρχήν να σας μιλήσω για την πολυσχεδία, αυτή διαδικασία της καινοτομίας. Όπως γνωρίζετε, Έχουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα που βασίζονται στη διδασκαλία, μαθήματα και αξιολόγηση. Αυτά είναι τα, αυτοί είναι οι τρεις ε, βασικοί πυλώνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουμε και την, το όραμα του σχολείου και τις καινοτομίες ως προς τα παιδαγωγικά συστήματα και την τεχνολογία. Αν δούμε την παιδαγωγική, έχετε την εξατομίκευση, ε, εξατομίκευση ε, εκπαίδευσης, ε, παιδαγωγική, μαθήματα και περιεχόμενο μαθημάτων. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και επίσης υπάρχει και το εκπαιδευτικό σύστημα in and out. Έχετε και τις τεχνολογίες προσέγγιση ένα προς ένα, τηλεεκπαίδευση καθώς και ανοιχτούς, ανοιχτά μέσα που σχετίζονται και με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και πρόσβαση στους ε, υπολογιστές καθώς και αξιολόγηση της καινοτομίας. Υπάρχει και το cloud computing, προσβασιμότητα, ευρυζωνικό και ούτω καθεξής. Υπάρχει άλλη μία διάσταση που είναι η χώρη εκπαίδευσης, χώρη εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση σε όλες τις συνιστώσεις. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδοξο. Ε, έχω έχουν επέλθει πολύ μεγάλες αλλαγές. Έχουμε τους ε, καθηγητές που ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει σε πολλά σχολεία στην Ευρώπη. Αλλά οι μαθητές θα πρέπει να δείξουν τι έχουν μάθει, ε, δηλαδή να καθίσουν στα θρανία και να προβούν σε ε, να ακολουθήσουν εξετάσεις ε, μεμονωμένα και σε απομόνωση κατά κάποιο τρόπο. Αυτά είναι τα συστήματα αξιολόγησης. Στο προηγούμενο πάνελ έγινε λόγος για την παιδαγωγική διαδικασία και την τεχνολογία. Ποιο οδηγεί ποιο. Γίνεται αυτή η συζήτηση επί αλλά τώρα, αν ορίσουμε την παιδαγωγική διαδικασία και ενσωματώσετε και την τεχνολογία, τότε η εκμάθηση, η εκμάθηση θα είναι βαθύτερη και απλούστερη. Αυτό αφορά και τις αναδυόμενες ε, τεχνολογίες στα σχολεία. Πώς ε, θα μεταχειριστούμε τους μαθήτες και τους δασκάλους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεχνολογία σε συνάρτηση με τους δασκάλους. Μόνο οι δάσκαλοι μαζί με την τεχνολογία θα κάνουν τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία εκπαίδευση και δραστηριότητα καθώς και κατάρτιση των ε, καθηγητών. Τώρα, τι κάνουν ε, τι κάνει το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Σχολείων. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τα σχολεία, τους ε, δασκάλους, καθώς και τα Υπουργεία Παιδείας μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, εκπαίδευσης στις ψηφιακές κοινωνίες. Δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε στοιχεία και δεδομένα σε σχέση με τις βασικές πολιτικές και συστάσεις, να υποστηρίξουμε τα σχολεία και τους ε, ε, δασκάλους μέσω e-training και επίσης να υποστηρίξουμε αυτά τα δίκτυα σχολείων στα πλαίσια της ε, καινοτόμου διδασκαλίας και προσεγγίσεων εκμάθησης. Η DigiConnect μας ε, ζήτησε μία μελέτη στα πλαίσια των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών μέσα στα πλαίσια του Erasmus Plus για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ως προς τις δραστηριότητες για να υποστηρίξουμε τα σχολεία, εμείς εξ ονόματος της Επιτροπής ε, έχουμε ε, τρία δίκτυα με 600.000 δασκόλους, δασκάλους, 2 εκατομμύρια ε, μαθητές. Η Γενική Διεύθυνση ε, Έρευνας προς προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη διαδικασία μέσω και των ε, STEM και του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη δικτύωση. Η τρίτη διάσταση είναι αυτό που ανέφερε και η πρό... πρόεδρος, δηλαδή στη... στις μελλοντικές αίθουσες διδασκαλίας. Εμείς ε, ε, δημιουργήσαμε ένα ε, εργαστήριο τάξης, Class Lab, όπου ζητούμε από τους καθηγητές να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία συνύπαρξης παιδαγωγικής και τεχνολογίας. Αυτό το σύστημα εξελίσσεται. Έχουμε 30 με 40 εργαστήρια ανά την Ευρώπη και έχουμε και τους, τους λεγόμενους πρέσβεις διδασκαλίας. Φυσικά η κατάρτιση δεν αρκεί για να προσελκύσουμε τους δασκάλους ε, στις, ε, ε, στην, στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και προσπαθούμε να προωθήσουμε μαθήματα μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Πέρσι είχαμε την 20η επέτειο αυτού του δικτύου και προσπαθήσαμε να ορίσουμε τους 10 τομείς όπου θα πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτό που μας απασχολεί είναι η δεξιότητες στο χώρο εργασίας, η κωδικοποίηση, η εκμάθηση. Ο δεύτερος ε, τομέας αφορά τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και ε, ο τρίτος τομέας αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες και ε, δικτύωση των σχολείων μέσα στα πλαίσια της επίσημης και ανεπίσημης διδασκαλίας που προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις για να προωθήσουμε και την καινοτομία. Και σε σχέση με το προηγούμενο πάνελ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά μέσα, το selfie και οι, οι ψηφιακοί, ψηφιακές αρμοδιότητες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η πλαισίωση αυτών των ε, μέσων έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την εργαλειοθήκη και για τους δασκάλους ε, και τους μαθητές. Ως προς τις, τις τέσσερις προτεραιότητες θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους μαθητές έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες σε μια ψηφιακή κοινωνία. Αυτό αφορά και τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την εκπαίδευση γενικότερα. Ε, γίνεται λόγος και για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ε, προσμιγνύουμε τα πάντα. Χρειαζόμαστε επαγγελματίες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ICT, και επίσης να έχουμε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού για όλους τους νέους και γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφορετικά μέσα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι δύο προκλήσεις δεν μπορούν να επιληθούν ε, ως εκμαγείας. Ο δεύτερος τομέας είναι να βοηθήσουμε το ε, προσωπικό των δασκάλων να έχουν να οικοδομήσουν τις ικανότητες τους και αυτό αφορά και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Η τρίτη διάσταση είναι τα, το νέο περιβάλλον εκμάθησης, τα νέα αυτά περιβάλλοντα για να υπάρχουν συνεργατικοί φορείς τους οποίους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί η τεχνολογία μας υποστηρίζει, αλλά πολλά επισυμβαίνουν. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι επίσημες και οι ενεπίσημες δυνατότητες να συνδέσουμε το σχολείο με μια ευρύτερη κοινότητα. Το είδαμε και μέσω STEM. Δεν υπάρχουν καθηγητές σε επίπεδο STEM στην Ευρώπη. Ε, ως προσθετικές δηλαδή επιστήμες. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτές οι, αυτοί οι νέοι χώροι ευελιξίας και επίσης η διαβάθμιση της ε, καινοτομίας. Ε, έχουμε πολλά πιλωτικά σχέδια σε πολλές χώρες. Προσπαθούμε να ε, έχουμε τη συμμετοχή πολλών σχολείων, έχουμε 4.000 σχολεία και το βασικό ζήτημα δεν είναι να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα, αλλά τη διαδικασία που οδήγησε στα αποτελέσματα. Τέλος, και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, η ε, ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει μία ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις επαγγελματικές πρακτικές σε επίπεδο σχολείου, έτσι ώστε να έχουμε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ICT, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και επίσης ένα δεύτερο στοιχείο είναι να αγκαλιάσουμε αυτή την ψηφιακή μετάβαση σαν αναπόσπαστο ε, ε, σημείο των σχολείων και να διαφωτίσουμε την όλη διαδικασία, να ρίξουμε φως στην ε, διαδικασία και στις πρακτικές διδασκαλίας και να έχουμε νέα στοιχεία για την έρευνα, να έχουμε νέα κριτήρια ε, αποτίμησης, να υπάρχει ε, εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα και επίσης να μπούμε σε μια διαδικασία περισυλλογής ε, στην έρευνα και φυσικά να ξανανακαλύψουμε την χαρά της διδασκαλίας. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη αυτή παρουσίαση θα προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους ομιλητές και θα το συζητήσουμε. Θα καλωσορίσω την Ιλώνα Κις, είναι υπεύθυνη του Δήματος, ε, διαβάζω και γράφω, για τις δημόσιες βιβλιοθήκες εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζουμε ότι οι βιβλιοθήκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψηφιοποίηση και γι' αυτό θα θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα από την κυρία Κίσα Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σήμερα και που συμπεριλαμβάνετε και τη βιβλιοθήκη σε αυτή τη συζήτηση. Το όνομα μου είναι Ηλώνα και εργάζομαι σε ένα πρόγραμμα εδώ στις Βραξέλλες για τις δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι ότι ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών στην ε, ψηφιακή εκπαίδευση και συγκεκριμένα στον αλφαβητισμό τις κριτικές δεξιότητες για τα βασι... τις βασικές ουσιαστικά ψηφιακές δεξιότητες για ανθρώπους που μπορεί να μην στην εκπαίδευση ή στην εργασία και το ρόλο που παίζουν οι δημόσιες Θα δούμε τις διάφορες εκθέσεις που έχουν αναφερθεί, το σχέδιο δράσης και συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη μεγαλύτερη έμφαση στην άτυπη μη τυπική εκπαίδευση στι ευρωπαϊκέ πολιτικές ώστε να συμπληρωθεί ε, ο διάλογος για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε τις στατιστικές. Είναι αξιοσημείο ότι ακόμα μέχρι σήμερα ένα μέσο όρος του 5% των πολιτών δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και αυτό αφορά άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή ε, ή το ίντερνετ, δεν ξέρουν πώς να ε, κάνουν ε, πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και αυτός είναι ο πληθυσμός για τον οποίο οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι χρήσιμες. Πώς άλλαξαν οι βιβλιοθήκες τα τελευταία 20 χρόνια. Είπατε ότι όταν πάμε σε μια τάξη σήμερα είναι σαν αυτή που πηγαίνετε όταν παιδί. Αυτό μπορεί να ισχύει και για αρκετέ δημόσιε στην Ευρώπη, αν και κάποιε αλλάζουν δραματικά. Υπάρχουν 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση και ε, εκεί μπορούν να δανειστούν βιβλία. Πάνω από 100.000 επισκέπτονται τις δημόσιες βιβλιοθήκες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια επανάσταση φυσικά στι υπηρεσίε που παρέχουν και στον τρόπο που λειτουργούν. Οι εικόνε που χρησιμοποιώ στην παρουσίαση έχουν τραβηχτεί από την ομάδα μας σε διάφορες βιβλιοθήκες ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση από τους ε, επισκέπτες των βιβλιοθηκών για βοήθεια σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες Έχουμε δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια, αλλά θεωρούμε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στι βιβλιοθήκε στην Ευρώπη. Θα θέλουμε να έχουμε και συγκρίσιμα δεδομένα από την υπόλοιπη Ευρώπη, να δούμε πόσα τέτοιου είδου αιτήματα λαμβάνουν οι βιβλιοθηκάρια από του επισκέπτε. Τέτοιε υπηρεσίε ζητάνε οι επισκέπτε. Ε, Μεγάλε βιβλιοθήκε έχουν ειδικά σημεία που μπορεί να έρθει κανεί και να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά αυτό είναι μια μεγάλη πρόσκληση του βιβλιοθηκάριου, γιατί θα χρειάζονται οι πόροι κατάλληλοι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ξενόμενες ανάγκες των επισκεπτών σε μικρές βιβλιοθήκες στην Υπέθρο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πού θα πάνε αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι ένας στους δέκα Ευρωπαίους έχει μηδενικό αλφαβητισμό και φυσικά και εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των πληθυκών στον βασικό αλφαβητισμό. Ψηφιακές δεξιότητες δεν αφορούν μόνο, δεν ε, ε, επηρεάζουν μόνο τους μεγαλύτερους ε, ανθρώπους Υπήρξαν πολύ πετυχημένα προγράμματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, για τη βοήθεια των μεταναστών, των προσφύγων, ε, για παιδιά που είχαν θέματα αλφαβητισμού. Ακόμα και σε ψηφιοποιημένες χώρες όπως είναι η Δανία, ακόμα και εκεί είναι πολύ σημαντικό το κοινό να μπορεί να κατανοήσει τα εργαλεία που έχει στα χέρια του και γι' αυτό... Ε, και πάλι ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι πολύ σημαντικός ο βιβλιοθηκάριος έχει έναν κεντρικό ρόλο και η βιβλιοθήκη παρέχει έναν ιδανικό σημείο συνάντησης όπου μπορεί κανείς να έχει ψηφιακές εμπειρίες και πολύ συχνά είναι το μοναδικό δημόσιο κτίριο στο οποίο μπορεί κανείς να μπει ελεύθερα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν ε, συσκευές κατάλληλες για πρόσβαση στο ίντερνετ. Θέλω να σας δείξω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι, είναι βιβλιοθήκη του Ελσίνκη που θα ανοίξει τις αρχές του Δεκεμβρίου και είναι ένα παράδειγμα μιας ε, φουτουριστικής σύγχρονης βιβλιοθήκης η οποία σχεδιάστηκε με 2.000 ιδέες των πολιτών του Ελσίνκη για το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες και αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να είναι σύγχρονες βιβλιοθήκες δεν είναι σκορισμένα μικρά δωμάτια με βιβλία. Είναι κάτι από το οποίο αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε. Για αυτήν την επιτροπή θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να μιλήσαμε με τον Επίτροπο και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για το Erasmus Plus. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι υπάρχει ενισχυμένη στήριξη στο πρόγραμμα αυτό. όμω χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα που θα στηρίξουν ε, την εκμάθηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό λείπει στις προτάσεις. Θα πρέπει να ξεκλειδώσουμε τα κοινωνικά ταμεία ώστε να είναι πιο προσβάσιμα για διάφορα τμήματα Ελπίζουμε αυτή η Επιτροπή και η επόμενη μετά τις εκλογές να συνεχίσει να ε, αποτελεί πρωταθλητή για την κοινότητα των βιβλιοθηκών. Θα τελειώσω με κάποιες εικόνες που σίγουρα πολλοί θα τις έχετε δει. Να σας θυμίσω ότι είναι βασική αξία για το ρόλο των βιβλιοθηκών να δίνει πρόσβαση στους πάντες με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών και των επισκεπτών. Αυτή είναι μια κεντρική αξία και είναι κάτι που θα πρέπει να στηρίξουμε. Κάναμε αναφορά στην εβδομάδα Code. Είναι η τρίτη χρονιά που θα έχουμε το Generation Code στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλω να σας προσκαλέσω και να δείτε παραδείγματα για το πώς λειτουργούν ε, οι βιβλιοθήκες στην Ευρώπη για να προωθήσουν τις ε, ψηφιακέ δεξιότητες και την πρόσβαση σε όλους. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει, σα ευχαριστώ πολύ. Η, προ... η σας ευχαριστώ πολύ για την ματιά που μας βοηθήσατε να ρίξουμε στον σημαντικό ρόλο των βιβλιοθηκών. Πριν ε, προχωρήσουμε στην συζήτηση, Απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό πρώτα στον κύριο Δομήνικο Γκάμπα Κόρτα από την Επιτροπή των Περιφερειών, ο οποίος και βέβαια ε, είναι ας πούμε το φυσικό επόμενο βήμα μετά από τον ρόλο των βιβλιοθηκών, ε, έρχεται να μιλήσει για την σημασία του τοπικού και του περιφερειακού επίπεδου και τον ρόλο των επίπεδων αυτών στην ψηφιακή εκπαίδευση. Είστε ο εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειών για το σχέδιο δράσεως για την ψηφιακή ε, παιδεία. Και ε, αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σας κύριε Γάμπα Κόρτα. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά κύριε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως ε, την πρόεδρό σας κυρία Κάμερ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την πρόσκληση, όπως είπα, γιατί στην Επιτροπή Περιφερειών θα εγκρίνουμε το πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Η κυρία Κώστα είχε συμμετάσχει στις εργασίες μας. Το πρόγραμμα δράσης έχει ως εξής. Εμείς ως Επιτροπή των Περιφερειών αρχίσαμε να εργαζόμαστε τον Μάρτιο και πρόκειται για μία γνωμοδότηση ύψης της σημασίας για τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες, δήμαρχους και ούτω καθεξής και τοπικούς φορείς από την ε, Μπολόνια ξεκινήσαμε με αυτή τη διαδικασία όπου τονίσαμε την σημασία της διδασκαλίας, την ε, ελευθερία του λόγου, την ανοχή, την ελευθερία της έρευνας, την ελεύθερη διακίνηση των ε, φοιτητών και ούτω καθεξής. Σε αυτή την γνωμοδότηση, η οποία είναι σχηνοτενής, θα τονίσω ορισμένα μόνο σημεία. Μιλάμε για συνετή χρήση των ε, ψηφιακών πόρων. Υπάρχει η διαδικασία ε, bullying, εκφοβισμού, ε, sexting, sextortion και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει ένα στρεσογόνος ε, παράγοντας στην διαδικασία αυτή και υπάρχει και ο φόβος του να παραμείνει κανείς εκτός. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προετοιμάσουμε τα παιδιά έτσι ώστε να έχουν κριτική σκέψη. Φυσικά ο, ο μεγάλος κίνδυνος και ανησυχία είναι ο, ο εξής. Πολλές φορές το διδακτικό προσωπικό χρειάζεται, χρήζει ειδική κατάρτισης έτσι ώστε να έχουμε μία νέα μεθοδολογία επεξεργασίας ε, δεδομένων. Επίσης χρειάζεται και η, η παροχή δωρεάν ε, υλικού, ψηφιακού υλικού, πέρα από τη, τα πνευματικά δικαιώματα. Όμως η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει σε επίπεδο περιφερειών είναι ότι υπάρχει μεγάλο ψηφιακό χάσμα που αφορά συγκεκριμένες ε, γεωγραφικές ε, περιφέρειες, ο νότος της Ιταλίας, ας πούμε σε σχέση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μεγάλο ψηφιακό χάσμα και φυσικά και χαμηλή συμμετοχή των γυναικών ιδιαίτερα σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές. Εντάχει λοιπόν υπάρχει και το θέμα των ε, πόρων και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το σχέδιο, πολιετές σχέδιο ψηφιακής εκπαίδευσης, δηλαδή πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, θα πρέπει να προωθηθεί η συνδεσιμότητα και η συνέργεια των υποδομών. Η Επιτροπή Περιφερειών θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε όλα τα επίπεδα. Επ' αυτού θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ειδική περίπτωση που αφορά την καμπανία, τη δική μου περιφέρεια που δεν αφορά μόνο την Νάπολη, αλλά 5 εκατομμύρια πολίτες σε σχέση με τη Λομβαρδία. Ε, πρόσφατα στην καμπανία χρησιμοποιώντας πόρους από το ΕΚΤ μαζί με το βασικότερο πανεπιστήμιο, το Φεντερίκο Σεκόντο, της περιοχής της Νότιας Ιταλίας του Τζόρνο προώθησε αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, όπου εκατοντάδες νέοι και απόφοιτοι και πτυχιούχοι ασχολούνται με τις εφαρμογές που ε, υπάρχουν στα πλαίσια νέου λογισμικού και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και για την δημιουργικότητα και την ε, συνεργασία. Έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πρωταγωνιστές και στο επιχειρηματικό πεδίο. Αυτό το πρόγραμμα ε, είναι ανοιχτό όχι μόνο στους ε, Ιταλούς φοιτητές, αλλά ε, προέρχονται πολλοί φοιτητές προέρχονται από τη Μεσόγειο έτσι ώστε να υπάρχει μία συμμετοχική διαδικασία. Είναι μία μέθοδος συνεργατική όπου οι επιχειρήσεις, οι φοιτητές αλλά και οι διδάσκοντες συμμετέχουν σε αυτή την ακαδημία και έτσι προωθούν δράσεις και όλα αυτά γίνονται στα αγγλικά. Έχουμε πολλούς νέους οι οποίοι έχουν μία νέα προσέγγιση εκπαίδευσης και προσεγγίζουν και τον χώρο της εργασίας. Υπάρχουν και θέματα προγραμματισμού των ε, διαφόρων σημείων διεπαφής, interface και ο τρόπος διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Πώς ε, προωθείται το θέμα του ε, επιχειρηματικού ε, προγραμματισμού. Αυτό δεν το λέω επειδή είμαι τοπικιστής, αλλά γιατί θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι πολύ συχνά ε, αμφισβητείται το ΕΚΤ και οι δαπάνες του. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι οι επιχειρήσεις και η περιοχή της Καμπανίας φτάσαν σε μια πολύ σημαντική εμπειρία. Μπορείτε να δείτε και το ε, Development Academy που είναι η ιστοσελίδα μας και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την επιτυχή ε, συνεργασία στην ε, περιοχή της Νότιας Ιταλίας και ελπίζουμε αυτή να είναι και η προσέγγιση για την προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών στα πλαίσια της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Θα προχωρήσουμε στην ε, συνήθη ε, διαδοχή ερωτήσεων-απαντήσεων, όπως εξήγησα πριν με τη διαδικασία ping-pong. Και μια και είναι εδώ, θα δώσω το λόγο αμέσως στην εισηγήτριά μας, κυρία Γιάννα Τούμ. Ε, αν θέλει Σα ευχαριστώ. Και πρώτα ζητώ συγγνώμη που ήρθα με κάποια καθυστέρηση γιατί ταυτόχρονα είχα άλλη ε, επιτροπή όπου παρουσίαζα μια έκθεση. Λίγα λόγια για την έκθεσή μου, αλλά κατάλαβα τώρα από αυτά που άκουσα ότι την έχετε συζητήσει ήδη. Πρόεδρος, την παρουσίαση τη εκθέσεως θα την κάνουμε αμέσως μετά. Πρώτα κάνουμε ένα γύρο συζητήσεων αν έχει κάποιε παρατηρήσεις για τα όσα μόλις λέχθηκαν ή αν θέλει να δεις μια ερώτηση στους πανελίστ, ε, ε, ήθελα να σου δώσω το προβάδισμα ως ε, εισηγήτρια. Στην έκθεσή σου θα έρθουμε ευθύ αμέσω. Στη διάρκεια τη επεξεργασία τη εκθέσεω, συναντήθηκα με πολλούς από διάφορες γενικές διευθύνσεις και άλλες επιτροπές και γνωρίζω τις τοποθετήσεις των μεν και των δε. Οι ερωτήσεις μου και οι παρατηρήσεις μου περιλαμβάνονται ήδη στην έκθεση. Σας ευχαριστώ όμως που ήρθατε. Ευχαριστώ για τις εισρωές ε, με τις οποίες συμβάλλατε και είναι κρίσιμο. Αν πάει κανείς στο σχολείο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Εγώ δεν ήξερα τα πράγματα αυτά. Έχουμε μεγάλο αριθμό σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν καν σύνδεση με το διαδίκτυο. Ούτε καν σύνδεση με το διαδίκτυο. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη και ε, προβήκαμε και στην ανταλλαγή απόψεων με τους κοιόδης συγητές ήδη πριν αρχίσω να συντάσω την έκθεση και συμφωνήσαμε όλες και όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες, συμφωνήσαμε ε, σχετικά με το γεγονός ότι το ποσό της ψηφιακής γνώσης στο μέλλον ή εν πάση περιπτώσει ήδη τώρα, πάντως σίγουρα στο μέλλον, θα αποτελέσει ε, την βάση για το νέο κοινωνικό χάσμα Δηλαδή ανάμεσα στου ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν, δεν θέλουν να μάθουν και να χρησιμοποιούν τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευέ, θα είναι τελικώς οι χαμένοι στην αγορά εργασίας. Αυτό για μένα είναι απόλυτα σαφέ. Και ίσως θα χρειαστεί να συζητήσουμε τέτοια πράγματα και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Άλλο ε, θέμα αυτό. Αυτό το υπόδειγμα μέσα στο οποίο ε, μεγάλωσα. Η μάνα μου μου είπε όχι θα πρέπει να διαβάζεις, να πάρεις το δίπλωμά σου και μετά θα ασκήσει ένα επάγγελμα μέχρι να πεθάνει. Αυτά τα πράγματα τελείωσαν, δεν θα ξαναγίνουν. Τελείωσαν ποτέ. Σω ούτε καν εγώ που είμαι ήδη 52 ετών. Και μιλούμε για του νεότερους τώρα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε, να μετασχηματίσουμε το υπόδειγμα αυτό ή το παράδειγμα αυτό και να τα λέμε αυτά μέχρι ότι όλοι τα κατανοήσουν. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, εγώ δεν άκουσα καμιά ερώτηση προς τους ειδικού, αλλά ίσως παρόλα αυτά θέλουν να τοποθετηθούν. Κύριε Ντουράντο. Ε, όπως είπα, ε, κάνουμε ένα γύρο ερωταποκρίσεων. Αν θέλετε όμως, αν δεν θέλετε να τοποθετηθείτε, δεν πειράζει. Είπατε, λέει ο κ. Ντουράντο, για την διασύνδεση των σχολείων με το διαδίκτυο. Να είμαστε όμως και προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι ένα σχολείο έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, ότι χρησιμοποιεί στη διδασκαλία. Υπάρχει θέμα υποδομών λοιπόν, ασφαλέστατα. Συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και την ε, σύνδεση με το ευρύ φάσμα και υπάρχουν πολλές σχετικές πρωτοβουλίες, ε, η Voucher Initiative, Wi-Fi για τα σχολεία και άλλα σχετικά πολλοί δήμοι ε, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξοπλιστούν τα σχολεία. Η δεύτερη πρόκληση όμως είναι γύρω από το θέμα πώς χρησιμοποιείται το διαδίκτυο στην σχολική διδασκαλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η εκπρόσωπος των βιβλιοθηκών. Σας ευχαριστώ. Μιλήσαμε πριν για ε, ψηφιακή ισότητα. Εγώ εννοώ ε, ισότητα στις ευκαιρίες και οι οικονομικές ευκαιρίες όπου πάλι αυτές υποσκάπτονται από την ψηφιακή ανισότητα. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών λοιπόν, λοιπόν οι οποίοι ε, λαμβάνουν ψηφιακή εκπαίδευση και άλλοι όχι. Πρόκειται για ε, δημοκρατική συμμετοχή εν τέλει, για την συμμετοχή στις εκλογές. Για... Δηλαδή μπορεί κανείς να κάνει τη φορολογική, τη ε, του δήλωση ε, επιγραμμικά μπορεί να παραγγείλει ας πούμε, διάφορα είδη επιγραμμικά. Ε, η, ψηφιακή τεχνολογία που μπαίνει στη ζωή μας διευρύνει το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν και να συμμετάσχουν επομένως στο κοινωνικό γίγνεσθε και αυτούς που δεν μπορούν. Και όσοι ε, τώρα παλεύουν και παλεύουν θα συνεχίσουν να παλεύουν και όλο και περισσότερο. Το ζήτημα της ε, ψηφιακή δεξιότητα είναι όντως και ζήτημα κοινωνικής συμμετοχής και όλο και περισσότερο. Δηλαδή με, ποια, με ποιον τρόπο θα μπορεί κανείς να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και εδώ χρειάζεται να προσέξουμε η ψαλίδα να μην ανοίξει υπερβολικά. Η κυρία Κώστα. Εντάχει, μία ερώτηση προς τους ε, τρεις. αυτό το ε, δίκτυο των ευρωπαϊκών σχολείων ξέρω ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία 10 χρόνων από τους υπουργού Εκπαίδευσης Σουηδίας και Ιταλίας. Είσαστε λοιπόν μία πλατφόρμα που επιτρέπει την μεταφορά διαδικασιών και την ε, κινητικότητα ε, του διδακτικού προσωπικού. Δημιουργήσατε και αυτή την ακαδημία που νομίζω ότι έχει μακρά πείρα και όπου συμμετέχουν ε, διδάσκοντες από 36 χώρες. Αυτή η Ακαδημία δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί έτσι ώστε να υπάρχουν περαιτέρω επενδύσεις από το ε, πρόγραμμα ψηφιακής ε, δράσης. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα όπου επενδύει πραγματικά η Επιτροπή. Σήμερα, ε, θεωρώ ότι οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις ε, περιφέρειες. Εσείς μιλήσατε για τη δυνατότητα χρήσης του ΕΚΤ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω. Υπάρχουν δυσκολίες και κάτι το τελευταίο. Φυσικά και εμείς ε, ήμασταν πολύ ε, ε, υπερήφανοι για αυτή την πρωτοβουλία της ε, καμπανίας και θα δούμε ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και στην Νάπολη αλλά και αλλού με βάση τις δράσεις αυτής της Ακαδημίας. Συμμετείχαν τουλάχιστον 100 παιδιά είναι η μόνη ακαδημία που δημιουργήθηκε από την Apple, από τα πανεπιστήμια και από τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα θέλαμε να ε, διευρυνθεί και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας που θα πρέπει να μεταφερθεί κι αλλού. Σας ευχαριστώ εσείς κύριε Ντουράντο. Φυσικά, όταν αναφέρετε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πιστή στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία, φυσικά και να καλοδεχούμενη τέτοιου είδου στήριξη είναι μια υπόσχεση των ε, Υπουργείων Εκπαίδευσης πριν από κάποια χρόνια και είναι η προσπάθεια των Υπουργείων να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε ήδη 22.000 δασκάλους ε, στην Ευρώπη από τις νότιες χώρες, άρα η γεωγραφική ισορροπία δεν ε, υπάρχει, δεν υπάρχει καλή κατανομή και προς το παρόν μπορούμε μονάχα να παρέχουμε μαθήματα μόνο στα αγγλικά. Αυτό δυσκολεύει τους δασκάλους που δεν ε, είναι τόσο καλοί στα αγγλικά και αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε να ενταχθούν σε ένα εθνικό πλαίσιο τα μαθήματα αυτά και να παρέχουν ε, ουσιαστικά και κάποιο είδου πιστοποίηση, ευρωπαϊκή πιστοσύνη που σε αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις ακαδημίες. Φυσικά μελετάμε όλες τις ε, δυνατότητες ώστε να παρέχουν περισσότερη στήριξη. Ευχαριστώ κυρία Κίσ. Τι θα πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να αποφεληθούμε από την ύπαρξη των βουλευτικών. Και εσείς γελάτε και εμείς γελάμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχει μια νέα πρόταση. Θα πρέπει να εξορθολογιστεί, να είναι πιο σαφής. Όλα θα πρέπει να είναι πιο σαφή. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την είσοδο. Από τις τοπικές κυβερνήσεις εξαρτώνται οι βιβλιοθήκες. δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Έχει να κάνει με το πώς θα καταλάβουμε για το πώς θα λάβουμε τις πληροφορίες, πώς θα, πώς θα θέσουμε προτεραιότητες, πώς θα έχουμε πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Υπάρχει μια νέα πρόταση ε, στο πλαίσιο του ESF+, Plus, νομίζω, ναι. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να ξεκλειδώσουμε ε, τη δυνατότητα εκπαίδευση για του ε, βιβλιοθηκάρου. Είναι προτεραιότητα αυτό για εμά. Οι βιβλιοθήκε τώρα είναι κόμβοι τη κοινωνία με πολλαπλές υπηρεσίες προς το κοινό και η ψηφιακή εκπαίδευση είναι μία από αυτές. Δεν θέλουμε μικρή χρηματοδότηση από δεξιά και αριστερά. Ξέρουμε ότι δεν ε, ε, ε, εντάσσεται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αλλά θα ήταν ε, πολύ καλό να μπορέσει να υπάρξει μόχλευση για να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Βλέπω ότι υπάρχει γενικά ε, κατανόηση και συμπάθεια στην αίθουσα. Το θέμα να δούμε πώς μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα. Θα σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορούμε στο πλαίσιο του ΕΣΕΦ να το εντάξουμε. Αυτό έχουμε μια γνωμοδότηση και για το ΕΣΕΦ γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θέλουμε να κάνουμε κάτι γιατί οι βιβλιοθήκες παίζουν κεντρικό ρόλο και γιατί παράλληλα πολλές κοινότητες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις βιβλιοθήκες τους και να τις ε, εξοπλίσουν όπως θα ήταν απαραίτητο για να μπορούν να προωθούν και την ψηφιακή εκπαίδευση. Κάτι για το οποίο δεν ο κύριος ε, Ντουράντο, να προωθήσουν την έννοια του digital citizenship, του ψηφιακού πολίτη. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να παίξουν ένα ε, σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε πώς μπορούμε να λάβουν οι βιβλιοθήκες ε, μια άλλη μορφή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πέρα από το περιφερειακό και κρατικό επίπεδο. Ο λόγος στον κύριο Γαρακώτα. Ήθελα να πω ότι ως Επιτροπή Περιφερειών θα θέλαμε να ε, τονίσουμε τον ρόλο των τοπικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της εταιρικής ε, σχέσης ιδιωτικού ε, δημόσιου τομέα. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και γι' αυτό πιστεύω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν ε, και ε, θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη επιθετικότητα κατά των μικρών κοινοτήτων ε, ιδιαίτερα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτή την συνεργασία μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και της συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και φυσικά ε, αυτό που μας απασχολεί είναι το μεγάλο ψηφιακό χάσμα. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση των διδασκόντων, διότι ένα παιδί έξι χρονών θα μπορούσε να έχει έναν δάσκαλο ο οποίος δυστυχώς δεν έχει ε, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και αυτό το παιδί βρίσκεται σε δυσχερή θέση εναντί άλλων παιδιών που έχουν ένα πιο φωτισμένο δάσκαλο. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει και η κατάρτιση του, των διδασκόντων, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στα όρια της ε, συνταξιοδότησης, που έχουν λιγότερο ενθουσιασμό και λιγότερες δυνατότητες προσαρμογής στην ψηφιακή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε όμως ε, να πλήξουμε τα παιδιά που είναι μικρά, ζουν σε μια μικρή χώρα όπου ο δάσκαλος ε, δεν είναι ιδιαίτερα καλός σε τέτοια θέματα ψηφιακής κατάρτισης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τρύπελ. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις καθώς και τις απαντήσεις που δώσατε ήδη. Επανέρχομαι στην ανάγκη των βιβλιοθηκών ως ε, κέντρο για την τοπική κοινότητα και βέβαια για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Στο Άρχους πήγαμε και είδαμε μια θαυμάσια ε, βιβλιοθήκη που ήταν ένα πραγματικό community center, πολύ ανοιχτή, πολύ έτσι στραμμένη προς την παροχή υπηρεσιών ε, συμπεριληπτική ας πούμε έτσι και ανοιχτή και από την αρχιτεκτονική σκοπιά είδατε, ε, ε, είδα και την εικόνα που δείξατε από την ε, ωραία αυτή βιβλιοθήκη στο Ελσίν και νομίζω η σκανδιναβική αντίληψη, η σκανδιναβική νοοτροπία ας πούμε έχει αντιληφθεί τι χρειάζεται να γίνει. Ε, τα είδαμε και στην επίσκεψη στην Silicon Valley αλλά εμείς εδώ στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτές τις μεγάλες, πολύ μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις παίκτες στην ψηφιακή οικονομία. Για ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε εδώ ε, μέσα από το δημόσιο ε, τομέα. Παλαιότερα ζητούσε η φορολογική αρχή από την μητέρα μου να στέλνει την ε, φορολογική της δήλωση ψηφιακά, να δηλαδή αποβάλει δηλαδή τα έγγραφα σκαναρισμένα. Και η, η, γυναίκα αυτή ήταν αδύνατον, δεν είχε τη γνώση ούτε και την πρόσβαση και εξαρτιόταν λοιπόν από τη βοήθεια των παιδιών τη. Αυτό συγγείει και πάρα πολλού ηλικιωμένου. Ε, αυτά που είπε και για το ESF, η Πέτρα προηγουμένω, αλλά και άλλα προγράμματα, ε, εκπαιδευτικά προγράμματα, σε όλα αυτά πρέπει να περιλάβουμε και το τι σημαίνει η ψηφιακή επανάσταση, η οποία συμβαίνει και στο χώρο δουλειά και στην υγεία και στην κοινωνική συμμετοχή. Παντού δηλαδή δεν είναι μόνο ένα μέρος της κοινωνίας. Ε, ε, ε, αναπτύσσεται παντού. Θα ήθελα τώρα να έρθω στο θέμα του κ. Ντοράντο, διότι νομίζω ότι είναι πραγματικά κρίσιμο για την επιτυχία της προσπάθειας. Μιλήσατε για την αύξηση της χαρά στη μάθηση. Δηλαδή είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Και από την άλλη μεριά να αναζωογονήσει κανείς και την χαρά του διδάσκοντος. Χωρίς αυτά τα πράγματα, βεβαίω ε, καμιά φορά η μάθηση είναι και δύσκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να παραμείνει μια πηγή χαράς απόλαυσης και να συνδυάζεται ε, αυτή η απόλαυση εκατέρωθεν, γιατί αλλιώ είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την παρατήρηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο, κυρία Κάμερ Εύερτ. Θα θέλατε να πείτε κάτι, ας πούμε, καταληκτικά. Άλλες ερωτήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ε, ε, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα και να έρθουμε στην έκθεση της κυρίας Τούμ, ε, λέει πρόεδρος. Η κυρία Κίσ. Ευχαριστώ κυρία την κυρία Τρίπελ που έρθει στο θέμα αυτό. Πράγματι στο Άρχους ελήφθη ρητή απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες μέσω του δικτύου βιβλιοθηκών. Μια πραγματικά φωτισμένη απόφαση ε, ε, ο κόσμος πάει εκεί συνεχώς και είναι εξοπλισμένη η βιβλιοθήκη για να μπορεί να τους ε, βοηθεί. Ας πούμε, μπορούν να ζητήσουν να εκδοθεί το διαβατήριό τους μέσω του δικτύου της, βιβλιοθήκη. της βιβλιοθήκης. Να κάνουν την φορολογική του δηλώση κλπ. Και πραγματικά έχει ψηφιστεί και ως η καλύτερη βιβλιοθήκη της Ευρώπης. Και στο Ελσίνκι θα είναι θαυμάσια μια επίσκεψη, αν και βέβαια το Ελσίνκι το Δεκέμβριο ε, θα είναι λίγο δύσκολα από άψη καιρού εννοώ. Ο κύριος Ντουράντο. Μιλώ για τη σημασία της συμφιλίωσης της τυπικής, άτυπης και ε, ουσιαστικής ε, μάθησης. Ένα μέρος της εκπαίδευσης γίνεται και εκτός των ε, τείχων του σχολείου. Τελείως διαφορετική πρόκληση λοιπόν για να ανοίξει το σχολείο στην ε, κοινότητα που βρίσκεται, περιβάλλουσα κοινότητα. όπου μπορεί να συνδυαστεί η τυπική και η μη τυπική ε, εκπαίδευση για να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες κάθε πολίτου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ντουράντο, λέει πρόεδρος, τελειώνοντας ο κύριο Γκάμπα Κόρτα. Eh, Μπορούμε να πούμε εν κατακλείδη ότι οι νέοι θα πρέπει να κατανοήσουν, να κατανοήσουν ότι πρέπει να ε, ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία για να μπουν και στην αγορά εργασίας. Υπάρχει το θέμα της εγκατάλειψης του σχολείου, ιδιαίτερα ε, από, είτε από μαθητές που δεν τελειώνουν το Λύκειο, είτε από αυτούς που γράφονται στο Πανεπιστήμιο αλλά δεν το ολοκληρώνουν. Θα πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στο να ε, καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα στο μέτρο του δυνατού. Η μάθηση πάντα αποδίδει. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίσ, κύριε Ντουράντο, κύριε Γκαμπακόρτα για τη συμμετοχή σας ε, στον δεύτερο γύρο και βέβαια και τους προσκεκλημένους μας του πρώτου γύρου. Ήταν ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για κάποια φορά η συζήτηση του σημερινού απογεύματο. Ακούσαμε πολλές προτάσεις και σχετικά ε, με τις δημοσιονομικές ε, διαβουλεύσεις που θα διεξαγάγουμε, αλλά βέβαια και επίσης πολλές υποδείξεις για την έκθεση πρωτοβουλίας, για την παιδεία στην ψηφιακή εποχή, για το τι έχουν να κάνουν τα πράγματα αυτά με την ευρωπαϊκή πολιτική. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ, για την ε, συμμετοχή σας στη συζήτηση, για το παράθυρο που μας ανοίξατε στη σκέψη σας. Θα παραμείνουμε σε επαφή και πολύ ευχαρίστως να παραμείνετε ακόμη εδώ για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της εκθέσεως πρωτοβουλίας της κυρίας Τούμ για το εισηγήτρια για την έκθεση πρωτοβουλίας με τίτλο «Παιδεία στην ψηφιακή εποχή, προκλήσεις και διαπιστώσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική» ε, για να έχει τον λόγο για πέντε λεπτά για να προβεί στην παρουσίαση της εκθέσεως. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω καταρχήν τη γραμματεία για την υποστήριξη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Συναντήθηκα με πολύ ενδιαφερόμενα μέρη, άκουσα διάφορου ομιλητέ και ένα πράγμα ήταν σαφέ ότι η τεχνολογία προχωράει πολύ γρήγορα και μετασχηματίζει τι ζωέ μα πλήρω. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει φυσικά να προλάβουν τι εξελίξει. Δεν έχει μόνο να κάνει με δεξιότητε τη ψηφιακή, αλλά και την χρήση τη τεχνολογία ω ένα εργαλείο στην εκπαίδευση και για τον τρόπο που διδάσκουμε. Η κοινωνία και η αγορά εργασία έχουν αλλάξει. Η εκπαίδευση ήταν αρκετή για να μπορεί κάποιο να εισέλθει στην αγορά εργασία. Αυτό πλέον δεν ισχύει και ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στο ίδιο μοντέλο. Οι συνεχεί αλλαγέ ε, απαιτούν ε, νέες αλλαγές, ε, να μπορούν οι άνθρωποι να προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα είναι η τεχνολογία στο μέλλον. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους πάντες ώστε να μπορούν να μαθαίνουν γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια διαβίου προσέγγιση στην εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, ώστε να μάθουν τα παιδιά να μαθαίνουν. Είναι εύκολο να το πούμε περισσότερο από το να το πράξουμε. Πολύ σημαντικό είναι ο ρόλο των δασκάλων. Στον πυρήνα όμω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ κρατών μελών και για το πώ διδάσκονται τα ψηφιακά προσόντα και πώ διδάσκεται η τεχνολογία. Είναι σοκαριστικό ότι υπάρχουν ακόμα σχολεία τα οποία δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο και συμφωνώ φυσικά με αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Ντουράντο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στην ε, εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως στα σχόλια αυτά που αναφέρθηκα πριν δεν χρησιμοποιείται καν η τεχνολογία. Ίσως κάποιοι ε, να κάνουν ε, αναφορά στο θέμα του εθισμού. Ο εθισμός είναι αποτέλεσμα των χαμηλών ψυχικών δεξιτών των γονιών τους. Όλα τα παιδιά αγαπούν τα γλυκά, όμως Ποιο θα έδινε στα παιδιά του ένα φλιτζάνι με ζάχαρη κάθε μέρα. Αυτό έχει να κάνει με εμά, με του ενήλικε και πώ χρησιμοποιούμε τεχνολογία σωστά. Υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν είναι λοιπόν συνδεδεμένα παρά ε, την ύπαρξη προγραμμάτων και χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο γιατί αυτοί που υποφέρουν από αυτό είναι οι μαθητέ. Πέρα από το θέμα τη συνδεσιμότητα, το πρόγραμμα, υπάρχουν και άλλα προγράμματα όπω το σχέδιο δράση για την ψηφιακή εκπαίδευση που συζήτησαμε σήμερα, καθώ και άλλε ανταλλαγέ βελτίστων πρακτικών. Πολλέ γενικέ διευθύνσει ε, τη Επιτροπή ασχολούνται με την ψηφιακή εκπαίδευση, πως δεν υπάρχει μια ε, κεντρική προσέγγιση. Τα πάντα γίνονται σε θελοντική ε, βάση και πολλές φορές τα σχόλια από μόνο θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα ισχυρό κίνημα βάσης, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αν δεν θέσουμε στόχους, είναι πιθανόν πολλά σχολεία απλά να μην μπορέσουν να κάνουν τη μετάβαση και αν δεν υπάρχει στόχος να πετύχουμε ένα επίπεδο δεξιότητα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τότε δεν θα υπάρξει καν ε, ε, το κίνητρο για να πετύχουμε τους ε, στόχους αυτούς. Αυτό θα αυξήσει μόνο τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που ήδη είδαμε στο διάγραμμα που μα παρουσιάστηκε από, από την κυρία, από τη την κυρία Είναι κάτι που με σοκάρει. Είμαι από την Εστονία και πάντα κάνουμε λόγο για digital. Άρα ήταν σοκαριστικά αυτά που παρουσιάστηκαν. Φυσικά αυτό το χάσμα, τη διαφορά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε στρατηγικέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φτάνω στο τελικό σημείο ότι πέρα από τι γενικέ στρατηγικέ θα πρέπει να υπάρξει ένα καταλληλός τρόπο να μετρήσουμε τις ψηφιακέ δεξιότητε Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, τις ενότητες της πίζα για τη γλώσσα και για τα μαθηματικά. Όμω, για τι ψηφιακέ δεξιότητε δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε ποιες είναι απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Θα πρέπει άρα να υπάρξει ένα παρόμοιο τεστ και για τις ψυχικές δεξιότητες, για να δούμε και να αξιολογήσουμε ποιο επίπεδο έχουν τα παιδιά, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να αξιολογήσουμε την πρόοδο. Θα, ε, το SELF είναι ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης το οποίο όμως δεν είναι επαρκές. Είναι τόσο σημαντική η τεχνολογία στη ζωή μας, που είναι τόσο σημαντική όσο η ανάγνωση και η γραφή. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο πώς βλέπουμε την εκπαίδευση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας σε αυτό το πεδίο και να ακούσω τις ιδέες σας φυσικά. Και θεωρώ ότι οι σκιώδεις συζητητές θα έχουν πάνω κάτω τις ιδέες απόψη με μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περάσουμε στους σκιώδεις συζητητές είναι σημαντικό και πάλι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και να υπάρξει ενότητα. Κύριος Μάλινοφ, εκ μέρους του ΕΛΚ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Επιβεβαιώνω ότι υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της συγγήτρια και των σκιωδών συγγητών. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα έχουμε δύσκολο διάλογο, ούτε διαφορές οι δυσκολίες που έχουμε προκύπτουν ουσιαστικά από την πολυπλοκότητα του θέματος. Γι' αυτό δεν θα υπάρχουν ιδεολογικές διαφωνίες. Το δικό μου το πρόβλημα είναι ότι με τη γενική αίσθηση που έχω όταν προσεγγίσουμε το θέμα αυτό υπάρχει ε, ένα αίσθημα απόγνωσης και πανικού όχι σε σχέση με την Apple, το Facebook και την Αμερική, αλλά με κάτι που συμβαίνει, στην κοινωνία και για το οποίο έχουν καθυστερήσει πολλοί πολιτικοί, έχουν καθυστερήσει να το αντιμετωπίσουν, γιατί πολλοί είπαν ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δεν γνωρίζουμε οι πολιτικές αποφάσεις που κάνετε ε, δείχνουν γενική αίσθηση ότι τη στιγμή που εγκρίνουμε κάτι στο κοινοβούλιο είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό ότι θα είναι απαρχιωμένο μέσα στα επόμενα χρόνια και πάντα έχουμε την αίσθηση ότι κάποιο κάνει, τα, κάνει κάποια πράγματα καλύτερα από ότι εμεί. Δεν μιλάω για την Αμερική απαραίτητα, μιλάω για τους δυτικούς φόρου για τι επιχειρήσει. Ή αυτό που ονομάζουμε κρατική Έχω πάντα αυτή την αίσθηση λοιπόν όταν ε, ασχολούμαι θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Άρα προσπαθώ να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και το απευθύνω αυτό και στην Επιτροπή. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση προς την ε, ως προς τον ε, αλφαβητισμό, ψηφιακό αλφαβητισμό και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι κάτι που ενδεχομένως μας πονάει, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Κάτι πάνω στο οποίο επίσης εργάζομαι και χαίρομαι που συμπεριλήφθηκε είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι είναι η πρόκληση, η μεγάλη πρόσκληση, για να το πω πολύ έτσι ήπια, σε αυτό συμφωνούμε. Και κάτι ακόμα, ούτε επιχειρήσει, ούτε κανεί άλλο δεν θα το κάνει αυτό. Θα πρέπει όλο αυτό το θέμα με τι ψηφιακέ δεξιότητε να το αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε ψηφιακοί πολίτε. Δεν το κάνουμε για εμά. Έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, γιατί οι επιχειρήσει ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Αλλά το πώ θα συνδέσουμε την ψηφιακή ικανότητα με τη δημοκρατία, αυτό είναι δική δικό έργο. Οι τροπολογίες λοιπόν θα κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Λιάννα Ροντρίγκες, δύο λεπτά. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το προσχέδιο και θα ήθελα να πω σε γενικές γραμμές ότι αποτελεί αυτό το έγγραφο μία καλή ε, βάση εργασίας. Περνάμε στην ψηφιακή εποχή, έχουμε ήδη ε, περάσει σε αυτήν, γι' αυτό θα πρέπει να δεχτούμε αυτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή θα πρέπει να είναι η βάση εργασίας μας, της ρουτίνας μας, έτσι ώστε να δούμε πώς οι νέοι και τα παιδιά μας παίζουν, επικοινωνούν και μαθαίνουν. Οι νέες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές και μέσα στα πλαίσια της ε, ψηφιοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη στις παιδαγωγικές ε, πρακτικές και να ενταχθούν σε αυτές. Θα ήθελα να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού. Ως προς τις ε, ψηφιακές ικανότητες έχουν μεγάλη σημασία για τους νέους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία αναλογικότητας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να δημιουργήσουμε πιο υπεύθυνους πολίτες. Δεν πρόκειται για αυτό σκοπό, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει στην αποφυγή των κοινωνικών αποκλεισμών. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες και των ε, ίδιων των καθηγητών. Γιατί η παραδοσιακή κατάρτιση που βλέπουμε στα πανεπιστήμια δεν αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα Τροπέλ, ένα λεπτό θα προσπαθήσετε. Λοιπόν, θεωρώ ότι ακούσαμε πολλά σήμερα το απόγευμα και φοβάμαι ότι η αξιολόγηση του κύριου Μάλλον, ότι χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη ανάλυση να ξεκινήσουμε την ε, έκθεση ω προς αυτά που ακούσαμε σήμερα. Ε, είναι σωστή. Θα προτείνω τροπολογίες, αλλά πιστεύω θα βρούμε μια κοινή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν 20 δευτερόλεπτα μόνο η παρέμβασή σας. Ε, μιλάω εκ μέρους του κυρίου Συνατζότο που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεση που δίνει έμφαση όχι μόνο στα ωφέλη της ψηφιοποίηση, αλλά και τι προκλήσεις, μία από τις οποίες είναι ότι δεν όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι σε όλους οι χειρονάκτες έχουν ίδια πρόσβαση και είναι πιο ευάλωτη στην ε, αλλαγή αυτή. Φυσικά η διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντική, αλλά και για όλο το κοινό, στο σύνολό του, για να καταλάβει τη διαδικασία της ψηφιοποίηση ως κάτι που γίνεται μαζί με αυτούς και όχι σε αυτούς. Για να μπορέσουμε να μεταβούμε στην ε, ψηφική οικονομία του μέλλοντος. Κάνετε λόγο για την έλλειψη συνδεσιμότητας στα σχολεία, την ανάγκη να ε, επανεκπαιδευτούν οι εκπαιδευτική. Το κόστος είναι ένα θέμα εδώ, ε, γιατί είναι πολύ ψηλό, γιατί οι δεξιότητες ε, ε αυτές, για αυτές τις δεξιότητες υπάρχουν, ε, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Άρα θεωρώ ότι ανοιχτά προσβάσιμα μαθήματα διαδικτικά θα ήταν κατάλληλη λύση. Κάνετε λόγο για εξχρονισμένες τάξεις ε, είπατε ότι δεν υπάρχει διαφορά με το παρελθόν. Τα παιδιά μου σήμερα ε, επεξεργάζονται διαφορετικά τις πληροφορίες και έχουν άλλο ε, χρόνο ως προς την ε, προσοχή τους. Θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά σωστά. Και η αναφορά που έγινε στην διερευνητική μάθηση και σε δημιουργικέ μεθόδους. Όλα αυτά ε, συμπεριλαμβάνοντα αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρξουν καινοτόμε ε, μέθοδοι εκμάθησης που θα συμπεριλάβουν τις τεχνολογίες και φυσικά ε, οι θύνοντες ε, θα πρέπει να λάβουν ε, τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα. Θα πρέπει να αυξηθεί η γνώση, να υπάρξει ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για να διαδοθούν οι πρακτικέ. πρακτικές. Και τέλος, ε, ότι το να ε, αλλάξουμε την κλίμακα για να ε, προωθήσουμε την ψηφιοποίηση είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο... Θα θέλετε να θέσετε και την στην Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται, όχι, οπότε μπορούμε να περάσουμε και πάλι, εφόσον θέλει η Επιτροπή να πει κάτι, ο λόγος και πάλι στην συγγύτρια. Μάλλον όχι, η Επιτροπή. Καλωσορίζουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης και θα παρακολουθούμε ε, την εξέλιξη με τις τροπολογίες. Θα σας ε, απαντήσουμε αναλόγως. Όπως μας ζητάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννα, λόγω σε σένα και πάλι. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ τους χειρόδες συζητητές, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, την εκπρόσωπο της Επιτροπής, για την θετική διάθεση που έχετε. Να ζητήσω συγγνώμη αν υπήρξε αίσθηση ότι πανικοβάλλουμε, ότι με... βρίσκομαι σε απόγνωση. Θα σας δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Έχω πέντε παιδιά. Ο μεγαλύτερος μου γιος είναι 29. Ο μικρότερος μου είναι 12. Όταν συγκρίνω τα δύο νοσοκομεία που γέννησα τα δύο αυτά παιδιά με αυτήν την απόσταση ηλικίε, είναι σαν 100 χρόνια πριν. Το... Όμως η τάξη είναι η ίδια. Στο ίδιο σχολείο πηγαίνουν. Το 1973 είχαμε το Μαυροπίνακα, τα Θρανία και έναν βαρετό δάσκαλο. Και το ίδιο συνέβη και με τον μεγάλο μου γιο και με τον μικρό μου γιο και βλέπω τώρα τι εγγονέ μου και, εγγονές μου και φοβάμαι ότι θα έχουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Συνάδελφοι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πάντα κάνουμε λόγο για το υπόδειγμα του φιλανδικού σχολείου. Ούτε πίνακα, ούτε θερανία, ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, πειραματισμό. Αυτό δεν είναι βαρετό. Η μελέτη πρέπει να είναι διασκεδαστική και αν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω πραγματικά ήταν ε, το αποκορύφωμα αυτό που είπατε τη συζήτηση, ε, δηλαδή η ε, μάθηση πρέπει να έχει ενδιαφέρον και να έχει πλάκα, όχι βέβαια σε τέτοιε σχολικέ αίθουσες σαν αυτέ που περιγράψατε και που συχνά τι ζουν και τα παιδιά. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω ότι λαμβανόμαστε όλε και όλοι αυτό. Υπενθυμίζω προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 Ιανουαρίου στι 11 θα ψηφίσουμε στις 20 Νοεμβρίου και ελπίζουμε τον Δεκέμβριο να καταλήξει το έγγραφο έκθεση, δηλαδή στην Ολομέλεια, κάτι που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ακόμη. Άρα 28 Ενάτου στις 11 προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Ε, καλή επιτυχία στην περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου, στην εισηγήτρια και στους κοιόδης Το θέμα 8 τώρα ακολουθεί της ημερησίας ε, διατάξεως που είναι εξέταση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής με εισηγητή τον κύριο Ζντρογεύσκη. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η Δευτέρα Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου. Κύριε Ζντρογεύσκη, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ και πρώτα ευχαριστώ την κυρία Τούμ που βλέπω ότι βγαίνει από την αίθουσα για αυτά που είπε και, ε, και εκτός πρακτικών τώρα. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Τρούπελ η οποία ήταν επικεφαλής ε, της ε, αντιπροσωπείας μας που πήγε στο Σαν Φρανσίσκο και η επίσκεψη αυτή μας επέτρεψε να δούμε νέες τεχνολογίες που μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την εκπαίδευση. Θέλω να πω πραγματικά ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε η κυρία Τούμ και είναι και σημαντικό να δει κανεί ε, πόσο ταχύτατες είναι οι εξελίξεις. Σημαντικό ε, για να μην μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Τώρα, θέλω να σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εν προκειμένου να πω ότι η βιομηχανία πολιτισμού είναι από πιο σημαντικέ. και δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κανονισμός αναφέρεται μοναχά στην ιστορική πολιτιστική κληρονομιά, de facto όμως δεν υπάρχουν αναφορές στην δημιουργική βιομηχανία, βιομηχανία δημιουργίας, πολιτικής δημιουργίας, όπου όμως πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ε, δημιουργία, στην πολιτιστική δημιουργία, ε, δραστηριότητα κλπ. Βεβαίω με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αναφέρομαι στο άρθρο 167 παράγραφος 4 και και τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ένωσης και ε, βεβαίως είναι σαφές ότι ε, η Συνθήκη λέει καθαρά ότι η ε, Ένωση οφείλει να χρηματοδοτεί τέτοιε δραστηριότητε, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Μιλούμε για κανονισμό ο οποίο περιορίζεται ε, να ε, φύγει ακροθυγώ, αν μπορώ να πω τον πλεονασμό αυτό, το θέμα. Τώρα, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη, το Ταμείο Συνοχή, είναι ταμεία τα οποία πρέπει να διοχετεύουν κονδύλια και στον πολιτισμό. διότι αυτό αποτελεί εγγύηση για την περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. Αποτελεί δηλαδή εγγύηση για το μέλλον της βιομηχανίας δημιουργίας πολιτιστικού περιεχομένου. Διότι εκεί, που, εκεί θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες αυτές. Και έχω και κάτι άλλο να σας επισημάνω. Πρόκειται Πρόκειται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε νέους και ευρύτερους δείκτες. Ε, ιδίως δε για την πλήρωση των στόχων, ε, στους οποίους αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Τούμ. Ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη. Ακολουθούν οι σκιώδεις ηγητές. Ο κύριος Νέκοφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που στήριζε την προσέγγιση του να υπάρχει ε, μια μεγαλύτερη ορατότητα για το θέμα αυτό ε, στον τομέα του πολιτισμού. Συμφωνώ ε, με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θα αρχίσω με το θέμα του προϋπολογισμού ε, συνοχής. Α Εδώ και μερικά χρόνια έχει υποβαθμιστεί το Ταμείο Συνοχής και ε, δεν θα πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να επομιστούμε το βάρος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως προς τα, τις χρηματοδοτήσεις για τους πέντε βασικούς στόχους είναι πολύ καλή. Μία ευφιέστερη Ευρώπη, χαμηλότερη χρήση άνθρακα, ε, συνδεδεμένη Ευρώπη, κοινωνική Ευρώπη, μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα, καθώς και εγκύτητα με τους πολίτες και υποστήριξη των αστικών και περιφερειακών περιοχών καθώς και των ε, παρακτήων. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει και στο επόμενο πολιετές. Γι' αυτό η Επιτροπή είπε ότι οι δύο πρώτοι στόχοι θα χρηματοδοτηθούν ιδιαίτερα και θα υποβαθμιστούν οι επόμενοι τρεις. Πιστεύω ότι το κοινωνικό ο κοινωνικός πυλώνας θα πρέπει να έχει να τύχει χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα. Υπάρχει και μια άλλη αδυναμία που βλέπω στον κανονισμό σχετίζεται με τους δείκτες του κοινωνικού πυλώνα. Βασίζονται στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Δεν υπάρχει επαρκής ε, περιγραφή. Θα προτείνω λοιπόν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να τονίσω ότι το 10% των χρηματοδοτήσεων για τις περιφέρειες θα πρέπει να μας απασχολήσουμε στα πλαίσια της ε, δημογραφικής κρίσης για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε πιο αποφασιστικά. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω Πλήρω την πρόταση ότι το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να καλύπτει τον πολιτισμό και να δίνει περισσότερη ορατότητα και να κάνει δυνατές τις επενδύσεις και τις τεχνολογίες και οι δημιουργικέ ε, βιομηχανίε που ταλούν το 5% του GDP. Θα επανέλθω με το έρτημα για τον προπολογισμό όταν θα μιλήσει ο κύριος Νίκο. Έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι το πόσο του προπολισμού για τα διαφορετικά ταμεία και έχει να κάνει με το ποσό του, στο σύνολο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η εξυλλόγησή μου ότι είναι δυνατόν να κάνει μόνο με ίδιους πόρους και τα κράτη-μέλη θα ε, προσφέρουν περισσότερα χρήματα. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στο πόσο αντιμετωπίσουμε τα κράτη-μέλη μετά από το Silicon Valley είμαι ακόμα περισσότερο πεπισμένη ότι αυτή η ιδέα είναι σωστή και ότι θα πρέπει να πείσουμε τους συναδέλφους, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης της ψηφικής ατζέντας, θα χρησιμοποιούμε περισσότερα χρήματα στο ευρωπαϊκό προλογισμό και τελείως θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Και όσον αφορά στα στο τομέα τη συνοχή υπήρξαν ε, ανακοινώσει στην κοινωνική τηλεόραση ότι 300 εκατομμύρια των θεωρητικών ταμείων δεν μπορούν να ε, ε, επενδυθούν εξαιτία τη έλλειψη ε, χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση για αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να ανεβάσουμε τον προπολογισμό, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στι περιφέρειε και τότε έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Άρα με τις διαπραγματεύσεις του επερχόμενο πολιτισμοσυνομικό ε, πλαίσιο θα πρέπει να, ε, να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα. Λοιπόν, ο λόγος στην Επιτροπή θα θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το εισηγητή για τη γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης και τα μέλη για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Έχω ορισμένα σχόλια ίσονος σημασίας. Καταρχήν ο πολιτισμός παραμένει μία από τις προτεραιότητες της προτάσεις Επιτροπής. Ο Επίτροπός μου προσδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα και θα λάβω υπόψη τις ε, τροπολογίες που έχουν προταθεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με τις μεταγενέστερες τροπολογίες ότι αποτελούν μεγάλη, αποτελεί μεγάλη πρόκληση να πείσουμε κράτη-μέλη να προσθέσουν και άλλους δείκτες. Δεν έχει σημασία το μάκρος του καταλόγου, πάντα προσπαθεί κανείς να τον μειώσει. Γι' αυτό θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τέλος, σε σχέση με τη συνολική χρηματοδότηση, διαθεσιμότητα και προκλήσεις. Νομίζω ότι ένα από τα σημεία που τόνισε η Επιτροπή στη συνολική της προσέγγιση είναι να μειώσει το διοικητικό βάρος μέσα στα πλαίσια της επιτροπής κατάχυνσης της χρήσης των ταμείων, των πόρων των ταμείων. Υπάρχουν ορισμένες ε, λίγο ενοχλητικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Δηλαδή θα πρέπει να περάσουμε από το 1 συν 3 στο 1 συν 2 μέσα στα πλαίσια της όλης χρηματοδότησης, διότι το 1 συν 3 δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με τις εκκρεμούσες πληρωμές. Ο βαθμός εφαρμογής είναι πολύ αργός. Δεν μπορούμε να τον δεχτούμε και για την περίοδο 21-27 και είναι ένα από τα ζητήματα που προσπαθούμε να προτείνουμε με τις ε, βασικές μας προτάσεις. Συνεχίζουμε. Ε, μία παρατήρηση. ένα ή δύο σημαντικό στοιχείο, αλλά θέλω να μιλήσω και για άλλα δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Άλλοι δείκτες όπου η προτίμηση έχει να κάνει με τον πολιτισμό θα πρέπει να αυξάνει και την ευελιξία του προγράμματος και να μην δυσχεραίνει το όλο σύστημα. Γιατί αν έχουμε δείξει ότι ένα πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον, αυτό είναι κάτι καλό. Για να μην γίνει πιο βαρύ το σύστημα και κάτι ακόμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν κάνουμε λόγο για τον πολιτισμό, λαμβάνονται αρνητικές αποφάσεις, παραδείγματος χάρη. Από πλευρά πολιτική συνοχή δεν μπορούμε ε, τηθούν νέα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και πολλές χώρες έχουν αποσυρθεί από συγκεκριμένα project που θέλαν να χρηματοδοτήσουν τον πολιτισμό. Οι περιφέρειες στην πράξη αποχώρησαν από αυτά τα προγράμματα. Αυτή είναι η τάση και στο μέλλον το 5% του δημιουργικού τομέα θα μειωθεί περαιτέρω αν δεν επενδύσουμε σε αυτόν. Ευχαριστώ τη Χέλγα Τρουπέ. που εκπροσώπησε την αποστολή μας στο Σαν Φρανσίσκο και ήταν πολύ σημαντικό αυτά που είδαμε εκεί, τι μπορεί να κάνουν μπορεί να κάνει δημόσια χρηματοδότηση στο, στο κομμάτι της τεχνολογίας και πώς ε, επωφελήθηκε μερική από αυτό. Και τέλος, θα σας παρακαλέσω για νέε τροπολογίε. Θα παρουσιάσω και εγώ δικέ μου τροπολογίε και θα σα παρακαλώ να τι υποστηρίξετε. Αυτό όμω πρέπει να κάνουμε να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις επενδύσεις αν δεν αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που θα δημιουργηθούν. Ευχαριστώ πολύ και την συγκητήρια και, τον, και τους σκιώδεις ε, Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στις 3 η ώρα ε, οι τροπολογίες, 8 Νοεμβρίου ψηφοφορία στην Ολομέλεια αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, είναι πολύ στενό. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης και αυτή είναι η πρόταση ε, γνωμοδότησης θέσης προγράμματος Invest EU. Ο συνάδελφος Τζαμπάσκι είναι εισηγητής, δεν είναι όμως παρόν. Η Έμα θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα το πολύ πέντε λεπτά. Uh, thank you, madam. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη εξ το του κυρίου Τζαμπάρσκι. Άρχισε το αεροπλάνο του, αλλά μου δίνει τη ε, δυνατότητα να παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότης του Άγγελ. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλά διαρθρωτικά προβλήματα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συντονίσει αυτά τα θέματα, έτσι ώστε το εύση κόσμε και συνδέοντας την Ευρώπη να ε, φτάσουν σε αυτή την οικοδόμηση. Το EU Invest θα λάβει υπόψη το συμβουλευτικό κόμβο και το, την ιστοσελίδα και την πύλη Invest EU. Το Ταμείο EU e θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη συγχρηματοδότηση των εταίρων. Μιλάμε για 650 δις ε, ευρώ επιπρόσθετη χρηματοδότηση για το 2021-2027. Ένας άλλος τομέας είναι η συστηματική χρήση από τα κράτη έτσι ώστε να διαθέσουν το 5% των ε, κονδυλίων συνοχής και επίσης ε, θα προωθήσουν την κοινωνική τις κοινωνικές επενδύσεις, τις δεξιότητες, τον κοινωνικό τομέα τις, ε, και τις επενδύσεις ε, για την συνοχή. Μιλάμε για βιώσιμη και σωστή επένδυση, ενίσχυση των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και όσο αφορά τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εύρωστη ε, και σωστή διαχείριση, να λάβουμε υπόψη τους νέους, διότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους νέους για να ε, προσπαθήσουν να ανορθώσουν και την οικονομία μας. Ο Άγγελ θα ήθελε να, λάβει τα, να ακούσει τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους σκιώδεις συζητητές και ξεχνάμε τον Λίτζι Μόργανο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, αναγνώσασα. Ε, ως προς την ουσία του σχεδίου δεν μπορώ παρά να πω ότι υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις. Πιστεύω ότι πρώτα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πιο σωστή. Δηλαδή μιλάμε για τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, την υποστήριξη των ΑΜΕΑ, των ΑΜΕΑ και την υποστήριξη προσφύγων μεταναστών. Και επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που ήταν ανέλικτη ως προς την δημόσια χρηματοδότηση, θα πρέπει να ε, τονίσουμε τον τρίτο πυλώνα που είναι μη κερδοσκοπικός. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς της αγοράς ε, με βάση το Invest EU. Χαίρομαι διότι ο εισηγητής λαμβάνει υπόψη τις, ε, τους πολιτιστικούς οργανισμούς και ελπίζω να τονίσουμε τον, ε, την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και την ε, δημιουργική πολιτιστική κληρονομιά που δημιουργεί και ποιοτική εργασία και προβάλλει τον πολιτισμό ανά την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα. Σε γενικές γραμμές ε, υποστηρίζω την ορατότητα του δημιουργικού κλάδου. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα InvestEU θα θέσει τα πράγματα σε μια νέα βάση. Πάντα κάνουμε λόγο για επενδύσεις Άρα κάποιες φορές για μένα είναι περίεργο τρόπο, είναι περίεργος τρόπος που εργαζόμαστε. Ναι, φυσικά, ε, ακόμα και στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ε, και στο πρόγραμμα του Juncker θα ήθελα να μην κάνουμε πανεκκινήσεις πάντα, ε, ε κάνουμε πανεκκινήσεις αλλά να συνδέουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Μπίλντι. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε και τον κύριο Συγητή. Σύμφωνα με το ε, δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής InvestEU λέει στη βάση της επιτυχίας του σχεδίου Juncker. Εγώ φοβάμαι τα χειρότερα γιατί μέχρι τώρα η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών εργαλείων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν ελλειπής. Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2017 για το COSME-IN ήταν πολύ πιο ε, δεινή από αυτήν που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνω από το 40% των ισολογισμών, ε, των κονδυλίων μάλλον, είχαν δοθεί σε επιχειρήσεις που είχαν ε, ανάγκη από χρηματοδοτήσεις, δηλαδή πολύ χαμηλό, σύμφωνα και με το 43% του 2011. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή οι εγγύησεις αυτές δεν δίνονται επειδή υπήρχε ε, ε, πτώχευση. Ε, μας παρουσιάζουν τα προγράμματα, τα προγράμματα αυτά σαν πανάκια για να ενισχύσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να αναμένει κανείς ότι με το νέο ε, πρόγραμμα θα σηκώσουν πάλι τον πύχη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ε, μας πείθουν. Η πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ε, η κυρία Κώστα, όχι, όχι, με συγχωρείς, μια στιγμή, με συγχωρείς, με συγχωρείς, Σίλβια, μια στιγμή. Όχι άλλο και ο ε, ο κύριο Ζάμι Ντίμεχ, ο οποίο ε, είχε ζητήσει όμω πριν το λόγο από την κυρία Κώστα. Θα μιλήσω εξ ονόματος του δικού μας ε, ε του κυρίου Ζαγοράκη, ο οποίος κολλείεται σήμερα. Εξ ονόματος του λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ζαμπάσκη για την εργασία του και να σας ε, πω και ορισμένε θέσει της ομάδας μου. Συμφωνούμε με τις περισσότερες τροπολογίες του εισηγητού που απηχούν και τις δικές μας προτεραιότητες και στόχους ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς έχει ανάγκη να επενδύσει περισσότερο σε ανθρώπινο δυναμικό με την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως για τους νέους ανθρώπους και τους νέους επιχειρηματίες. Οφείλουμε ε, να εξασφαλίσουμε βιώσιμες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, να ενισχύσουμε έτσι την απασχόληση και την ανάπτυξη και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες. Όπως πολύ σωστά τόνισε και ο εισηγητής ή τονίζει μάλλον στο κείμενό του. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε περαιτέρω τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, παιδαγωγικά ιδρύματα και να δώσουμε και μικροχρηματοδοτήσεις. Να αντιμετωπίσουμε και σημαντικές κοινωνιακές προκλήσεις όπως τις δημογραφικές. Να ενισχύσουμε περισσότερο τους νέους και τη βιωσιμότητα, ιδίως τις ανάγκες νέων ανθρώπων σε νησιωτικές, ορεινές και υπαίθριες περιοχές. Να επενδύσουμε σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς. Εκεί όπου μπορεί να προσφέρει προς τη περισσότερη προστιθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ε, εγγυήσεις μέσω του προϋπολογισμού της. Δηλαδή, τις υποδομές, βιώσιμες υποδομές, έρευνα, ψηφιοποίηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές ε, δεξιότητες και είναι ρόλος μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσουμε περισσότερες επενδύσεις και συνέργειες στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην παιδεία και περισσότερα κονδύλια για τις σχετικές υποδομές ώστε να οδηγηθούμε σε τοπική ανάπτυξη ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο εισηγητής μας θα καταθέσει κάποιες τροπολογίες για να τονίσει τον ιδιαίτερο ρόλο των ε, τομέων αυτών και για να εκφράσει την ανησυχία του για την έλλειψη επενδύσεων σε θέματα ε, πολιτισμού, αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομίας. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, κυρία Κώστα, για ένα λεπτό σας παρακαλώ. Κάτι θα ήθελα να διευκρινίσω. Είναι τέσσερις ε, οι τομείς επενδύσεων στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα δεν αναφέρεται κάτι. Ε, και πέρα από τις ΜΜΕ θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική δικαιοσύνη, αρμοδιότητες και πολιτισμό. Και επειδή το Ταμείο Εγγυήσεων ε, εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να μιλήσουμε για μια δημιουργική Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό το Ταμείο, παρόλο που μπήκε στη ζωή μας δύο χρόνια πριν, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Οι ε, χρηματοδοτήσεις είναι 50% στον πολιτισμό και 50% στις ε, ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επενδύσεις και τις ικανότητες των φορέων. Και επίσης ε, να λάβουμε υπόψη και τους εμπειρογνώμονες, στο ρόλο των εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Σας ευχαριστώ. Ε, πάλι η ΕΜΑ, εξ ονόματος του εισηγητού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ανησυχίες σας, την υποστήριξή σας και φυσικά μας ενδιαφέρει το streamlining, η η και ενιαία πρόσβαση σε, αυτή, σε αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης που είναι ε, ύψης της σημασίας. Αλλά όλα αυτά θα τα αναφέρω στον κύριο Τζαμπάσκι και θα συνεργαστείτε μαζί του. 1η Οκτωβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ, Έμα, και εγώ θα το έλεγα αυτό. Προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών για το, 1 ε, ε, δεκάτου στι 5 το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στι 8 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Πολιτισμού και η Επιτροπή ΕΚΟΝ μαζί με του προπολογισμού θα ψηφίσουν στι 20 Νοεμβρίου. Και εδώ λοιπόν είναι ε, σφιχτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο καλούμε να τηρήσουμε. 1η Οκτωβρίου, 5 το απόγευμα για τι τροπολογίε. Σα Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος της ε, ημερησίας διατάξεως just in time ας πούμε. Θα ήθελα μόνο να σας επισημάνω ότι η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται στις 10 Οκτωβρίου 9 έως 12.30 και 3 έως 6 και 30. και στις 11 Οκτωβρίου 9 έως 12 και 30 και ελπίζω να σας δω όλες και όλους εδώ. Η κυρία Τρούπελ για ένα διάφορο. Μία ερώτηση για το AVMS την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Προβλέπετε μόνο ε, ψηφοφορία ή και συζήτηση. Πρόεδρος, νομίζω δεν θα διεξαχθεί συζήτηση παρά μόνο ψηφοφορία. Τουλάχιστον ο σχεδιασμός αυτό είναι ως τώρα. Διότι και εκεί είναι τόσο περιορισμένα χρονικά τα πράγματα ώστε να μην προλαβαίνει να γίνει τίποτε άλλο. Τουλάχιστον αυτό έχω πληροφορηθεί. Καλώς λοιπόν, σας ε, ελευθερώνω. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τις και τους διερμηνείς για την υποστήριξη του έργου τους. Ευχαριστώ.